αντιθουν με διερμηνείς ε, προβλέποντες συνεδριάσεις και ομάδες επισκεπτών την Πέμπτη θα, μπορούν ε, να, θα μπορούμε να τις υποδεχθούμε την Πέμπτη εδώ. Πρόεδρος, ε, ακούστε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της ερώτησής σας. Ενημερωτικά λοιπόν προετοιμάζω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα υπογράψω εγώ ίδιος ως πρόεδρος και θα απευθύνεται σε όλα τα μέλη. Σε όλους εσάς κυρίες και κύριοι ο καθένας που θέλει να έχει αυτές τις πληροφορίες θα πάρει αυτές τις πληροφορίες. Θα σας αποσταλεί αυτό το email, το ηλεκτρονικό μήνυμα γύρω στις 11 η ώρα και θα συμπεριλαμβάνει ακριβώς όλα τα στοιχεία τις απαντήσεις στις ερωτήσεις όπου γνωρίζουμε τις απαντήσεις. Μία από τις απαντήσεις είναι κάτι το οποίο μόλις ζητήσατε να πληροφορηθείτε. Την Πέμπτη λοιπόν όλες οι συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών ομάδων θα διεξαχθούν χωρίς ψηφοφορίες. Θα διεξαχθούν συνεδριάσεις αλλά χωρίς ψηφοφορίες περισσότερο θα έλεγα άτυπου χαρακτήρα τέτοιες συνεδριάσεις θα μπορούν να διεξαρθούν θα είναι εδώ παρόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά δεν θα γίνει ολομέλεια όλα λοιπόν τα άλλα εκτός ε, από τη διεξαγωγή της ε, Ολομέλειας ε, θα διεξαχθούν ομαλά, θα διεξαχθούν κανονικά. Επισκέπτες, ομάδες που θα προσέθουν στο Στρασβούργο να επισκεφθούν την Ευρωβουλή θα ε, τις υποδεχθούν όσοι, τους, ε, έχουν προσκαλέσει αυτές τις ομάδες θα έχουν πρόσβαση στα, στο κτίριο, θα μπορούν να προσέθουν και στην αίθουσα της Ολομέλειας, χωρίς όμως να διεξαχθεί η Ολομέλεια. Αυτή θα είναι η μόνη διαφορά. Δεν θα διεξαχθεί η Ολομέλεια, και δεν θα, γίνει και, δεν θα γίνουν και ψηφοφορίε στις ε, κοινοβουλευτικέ συνεδριάσει των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Διότι συμφωνήσαμε ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα διεξαχθεί καμιά ψηφοφορία. Όλα τα υπόλοιπα θα διεξαχθούν κανονικά ω εργασίε την Πέμπτη. Επαναλαμβάνω λοιπόν την Πέμπτη και Παρασκευή μπορείτε να υπογράψετε την, τον πίνακα παρουσιών. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό. Για την Πέμπτη και την Παρασκευή ο πίνακας παρουσιών, ο, ο κατάλογος θα είναι διαθέσιμος προς υπογραφή. Όλες οι επόμενες ε, ε, διαδοχικά πληροφορίες θα σας γνωστοποιηθούν στο ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα λάβετε και αυτό όχι αργότερα από το μεσημέρι πριν από το γεύμα. Θα γνωρίζετε λοιπόν τι θα έχει συμφωνηθεί σχετικά. Και χθε στην διάσκεψη των Προέδρων που έγινε και το Προεδρείο του Κοινοβουλίου συναντήθηκε και πολλά έχουν, ε, συμβαίνουν και συνέβησαν όσον αφορά τη σημερινή μέρα, από σήμερα θα αρχίσει να λειτουργεί μια ειδική ομάδα Task Force που θα συμπεριλαμβάνει υπηρεσίε του Κοινοβουλίου. Θα βρίσκεται διαρκώ σε επαφή μαζί μου αυτή η ειδική ομάδα και εγώ θα είμαι σε επαφή με του Προέδρου των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Πρέπει να υπάρχει διαρκή συνεχή ροή πληροφοριών σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν επιπτώσεις και αφορούν τις εργασίες μας και για αυτή την εβδομάδα και για τι επόμενε εβδομάδε. Να θυμάστε βέβαια την επόμενη εβδομάδα οι κοινοβουλευτικέ συνεδριάσει των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα διεξαχθούν, πρέπει να διεξαχθούν, δεν μπορούν να στροχοπεδηθούν, να σταματήσουν αυτέ οι εργασίε. Πρέπει να προπασκευαστούμε λοιπόν και για τι συζητήσει μα στις Βρυξέλλες. Δεν έχουν ληφθεί κάποιε αποφάσει ακόμα για αυτό το θέμα, όμω θα ληφθούν αποφάσει τι επόμενε ημέρε σε σχέση με αυτά τα θέματα. Μπορείτε λοιπόν να αναμένετε κάποιες σύντομες πληροφορίες από πλευράς μου, ενημέρωση όσον αφορά τις, ε, τις ε, τα, τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν στο άμεσο μέλλον. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση Τη ευρωπαϊκή επιτροπή και του Συμβουλίου όσον αφορά την διακοπή των συγκοινωνιών στην ενέργεια κυκλοφορία στην Ευρώπη. Εισαγωγικά θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Και καθώς γνωρίζετε, αποφάσεις που λαμβάνονται για τις επόμενες ε, ημέρες ε, θα πρέπει να ληφθούν από το εκτελεστικό σκέλος ε, των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Και φυσικά αυτό θα είναι έργο το οποίο θα αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν δραστηριοποιηθεί και δρούν από την προηγούμενη Κυριακή από κοινού. Εμείς όμως ως Ευρωβουλευτές έχουμε και εμείς κάποια καθήκοντα σχετικά και αυτά αφορούν μια μακροπρόθεσμη απάντηση, ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο που πρέπει να εξευρεθεί για να επιληθούν τα προβλήματα αυτή τη κρίση. Θέλουμε να εμπλακούν και οι, Ευρω... και οι κοινοβουλευτικέ μα επιτροπέ σε αυτό το εγχείρημα, να βρούμε πώ θα απαντήσουμε στα θέματα κατά τη διάρκεια της μήνυ ολομέλειας ε, στις Βρυξέλλες. Υπάρχει δυνατότητα μέσω ψηφίσματος, για παράδειγμα, να τοποθετηθούμε ή και να δράσουμε αντίστοιχα. Απευθύνω έκκληση λοιπόν σε εσά κυρίε και κύριοι να σημειώσετε επίσης ε, στις παρεμβάσεις σας πώς ε, ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συνεισφέρει για να επιληθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν για να μπορέσει κανείς να μετακινηθεί προς ε, το Στρασβούργο ή προς τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει όμως ε, να επικεντρωθούμε κυρίως στο πώς θα επιληθούν τα προβλήματα που αφορούν τους πολίτες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, έχουν πληγεί από αυτά τα προβλήματα σε σχέση με τις διαταραχές των ε, εναερίων μεταφορών. Να σκεφτείτε και να δείτε τι μπορούμε εμείς ως Ευρωβουλευτές να κάνουμε και να συνεισφέρουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τους πολίτες μας διότι στις αρχικές ώρες και ημέρες το κύριο βάρος των ευθυνών είναι του εκτελεστικού. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου για το ότι είναι παρόντες εδώ και θέλω να ζητήσω να ξεκινήσει το Συμβούλιο. Ίσως ο κύριος Γκαρίγκα θα μπορούσε να ξεκινήσει. Έχετε τον λόγο παρακαλώ κύριε Υπουργέ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουν όλοι, η εναέρια κυκλοφορία είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Αφορά τους πολίτες, την καθημερινή τους ε, ζωή, το, δικαίωμά τους, ε, το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και φυσικά αφορά και την οικονομική δραστηριότητα με αποφασιστικό τρόπο. Όταν λοιπόν οι εναέρειες κυκλοφορίες έχουν προβλήματα, όταν υπάρχουν στρεβλώσεις, και αυτό μάλιστα επηρεάζει πολλές χώρες και όχι μόνο μία. Διαφαίνεται σαφώς ο στρατηγικός χαρακτήρας αυτής, αυτού του μέσου και οι επιπτώσεις είναι πάμπολες. Και επειδή ακριβώς αυτή τη στιγμή το φαινόμενο επηρεάζει πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο, μία κρίση αναπάντεχη, μία κρίση χωρίς προηγούμενο, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Υπάρχει επίσης το παράδοξο ότι αντιμετωπίζουμε ένα θέμα στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει και τόσες αρμοδιότητες, έχει πολύ λιγότερες αρμοδιότητες από ό,τι σε άλλα θέματα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δράσει, θα πρέπει να αντιδράσει. Ενώπιον λοιπόν αυτή τη εναέρεια κρίση στην Ευρώπη, διαπιστώνουμε δύο πράγματα. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, ήταν πάρα πολύ σοβαρή κρίση, αλλά ταυτόχρονα είναι και ελάχιστο το επίπεδο ε, στο οποίο έχουμε νομικές δυνατότητες για άμεση δράση ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώ βρισκόμαστε ενώπιον μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούμε να κινηθούμε από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και αν αντιδράσαμε γρήγορα. Εδώ έγινε και το δεύτερο σημείο των σκέψεών μα. Τι κάναμε, πώ δράσαμε. Καταρχά, τα κράτη-μέλη, οι αρχέ ε, πολιτικής αεροπορίας εφάρμοσαν το υφιστάμενο πρωτόκολλο για τις επιπτώσεις ε, ηφαιστειακής τέφρας. Υπάρχει το Γραφείο ηφαιστειακών Επιπτώσεων στο Λονδίνο, το οποίο ασχολείται με τέτοια θέματα ε, και εφάρμοσε αμέσως τα όσα ε, αφορούν τους περιορισμούς της πτήσης και αυτό και έκανε ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και τους ελάχιστους δυνατούς κινδύνους για αυτή την πρώτη φάση δράσεις. Ε, είχαμε και δράση από πλευράς ε, Eurocontrol επί τη βάση των γνωμοδοτώσεων της επιστημονικής ε, ομάδος που υπάρχει στο Λονδίνο που έχει δημιουργηθεί εδώ και κάποια χρόνια και ασχολείται με την ηφαιστειακή τέφρα. τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα θεσμικά όργανα, άρχισαν να εργάζονται αμέσως και τις τελευταίες ημέρες είχαμε μια σειρά από τεχνικές συνεδριάσεις και τελικά καταλήξαμε στην χθεσινή απόφαση, η οποία ήταν πολιτικού χαρακτήρα από πλευράς Υπουργός Μεταφορών. Όλο το Σαββατοκύριακο ήμασταν επιποδός. Ε, η Ισπανική Προεδρία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως με τον Επίτροπο Κάλλας, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη διαθεσιμότητά του και για το χρόνο που διέθεσε, καθώς επίσης και με τη Eurocontrol, για να υπάρχει μια αντίδραση πολύ πιο συγκεκριμένη και θα είναι πιο κατάλληλα προσαρμοσμένη ώστε να μην έχουμε μια πιο μακροχρόνια κρίση η οποία μπορεί να έχει πάρα πολύ σοβαρέ επιπτώσεις για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωση και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από όλα αυτά λοιπόν προέκυψαν η σύσταση από πλευρά Eurocontrol, την οποία υιοθέτησαν ομόφωνα στη χθεσινή συνεδρίαση που έγινε με την Eurocontrol, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο αρχές ε, πολιτικής αεροπορίας, ε, ε, οργανώσεις εναέριας, εναέριων πτήσεων και όλοι συμφωνούν ότι από σήμερα θα πρέπει η Eurocontrol να καθορίσει τρεις περιοχές οι οποίες πλήττονται από την ηφαιστιακή πέτρα, τέφρα, συγγνώμη, μία ζώνη η οποία θα είναι η ζώνη στην οποία υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα τέφρας, εκεί θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση πτήσεων, μία δεύτερη ζώνη η οποία θα είναι εντελώς αντίθετο, δεν θα υπάρχει καμία παρουσία τέφρας και επομένως θα είναι ελεύθερη για πτήσεις και μία ενδιάμεση περιοχή στην οποία υπάρχει χαμηλή πυκνότητα τέφρας και θα επιτρέπεται να γίνονται πτήσεις χωρίς κίνδυνο και αυτή η περιοχή θα εξετάζεται με τα δεδομένα τα οποία δίνονται καθημερινά, κάθε έξι ώρες από πλευράς Eurocontrol και από εκεί και πέρα θα αποφασίζουν οι εθνικές αρχές συντονισμένα κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχουν αεροδιάδρομοι στους οποίους θα επιτρέπονται οι πτήσεις. Η σύσταση αυτή, η οποία προέκυψε από την ε, Eurocontrol, την οποία μας πρότεινε η Eurocontrol και είναι τεχνικού χαρακτήρα, έγινε δεκτή από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως θεωρούμε ότι είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα αυτό και προσπαθούμε να δούμε τι είναι απαραίτητο να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει απόφαση και από εκεί και πέρα προτείνει στα κράτη-μέλη να δράσουν. Υπάρχει λοιπόν μια ομόφωνη δέσμευση από πλευρά ε, ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει τη προτάσεω τη Eurocontrol για να δράσουμε. Θεωρήσαμε ότι η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια. Δεν υπάρχει κανένα συμβιβασμό από αυτού του θέματο, όπω είπε και ο Επίτροπο Κάλλα το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια περιοχή στην οποία υπάρχει δέσμευση να υπάρχει απόλυτη απαγόρευση πτήσεων. Ε, θα κάνουμε μια πολύ πιο ακριβή μελέτη της κατάστασης βάσει των δεδομένων που θα χρησιμοποιεί και η Eurocontrol, όχι μόνο δεδομένα τα οποία θα λάβουμε από τη Λονδίνα, αλλά θα υπάρχουν και δοκιμέ, οι οποίες θα γίνονται συνεχώς ε, από τις πτήσεις οι οποίες γίνονται δοκιμαστικά χωρίς επιβάτες. Ε, στοιχεία επίσης τα οποία θα λαμβάνουμε από τους κατασκευαστές των εξαρτημάτων των αεροπλάνων και από την υπηρεσία η οποία βρίσκεται στην ε, κολονία για να καθορίσουμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν αυτές οι τρεις περιοχές που συμφωνήθηκαν εχθές στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών. Ε, το οποίο συνεκάλεσε η Ισπανική Προεδρία. Πρόκειται λοιπόν για μια δουλειά η οποία θα είναι πολύ συντονισμένη, επί επιστημονικής βάσεως καταρχάς, θα βασίζεται και σε τεχνική απόφαση από τη Eurocontrol και σε μία απόφαση των κρατών μελών για αυτήν την ενδιάμεση περιοχή και εκεί θα πρέπει φυσικά να υπάρχει συντονισμός Εχθέ ήταν πάρα πολύ σαφής η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέσουν στους πολίτες και να κάνουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ό,τι άλλο μέσο εναλλακτικό μεταφοράς μπορούν να τους προσφέρουν για να αντιμετωπίσουν τις πολύ σοβαρές περιπτώσεις ε, μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών και των υπολείπων φυσικά πολιτών, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και φυσικά συζητήσαμε και τις πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης. Αυτά θα σας εξηγήσει ο Επίτροπος Κάλλας. Θα συστηθεί μια task force ε, Επικεφαλή θα είναι ο Αντιπρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπο Κάλλα. Θα συμμετέχουν και ο Επίτροπο Αλμούνια και ο Επίτροπο Όλη Ρεν. Και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει και η σχετική έκθεση, η οποία θα αφορά όλε τι οικονομικέ επιπτώσει. Τέλο, το συντομότερο δυνατόν, θα γίνει ένα νέο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών προκειμένου να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό ακριβώς, ε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια απόφαση για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προοπτική, ένα ευρωπαϊκό συντονισμό για όλα όσα συμβαίνουν, ε, λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τι αποφάσει για τι πτήσει, προστατεύοντα πάντα του πολίτε μα και χαίρομαι ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπούζεκ, ότι το γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μια συζήτηση ει βάθο του θέματο. Η συζήτηση αυτή σημαίνει ότι θα υπάρξουν σκέψει και ιδέε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, τα προβλήματα τα οποία πλήττουν τους λαούς της Ευρώπης και φυσικά μακροπρόθεσμα να δούμε τι δρέσεις πρέπει να αναλάβουμε ε, για αυτήν την αναπάντεχη και νέα κρίση η οποία όμως έχει πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες ε, τις επεξηγήσεις σας. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, διαβεβαιώσω και θα ήθελα να το διαβιβάσετε αυτό στην Ισπανική Προεδρία, στο Συμβούλιο Υπουργών, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευχαρίστω θα συνεργαστεί. Είμαστε έτοιμοι, ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση και στις επιτροπές ε, του ε, Κοινοβουλίου, οι οποίες εργάζονται ευχαρίστως ε, να συζητήσουμε με εκπροσώπους και της Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε εκλεγεί από πολλές ε, εκλογικές περιφέρειες ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη και επομένως είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε ό,τι μας επιτρέπεται νομοθετικά, δεν μπορούμε εκτελεστικώς να αναλάβουμε τίποτε, αλλά ευχαρίστως να συμμετέχουμε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα λάβει το λόγο ο Επίτροπος Σινκάλας. Για το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω την έκθεση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την ε, κρίση της εναέρειας κυκλοφορίας ε, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Ιλανδίας γνωρίζετε ότι χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και αυτό επηρεάζει χιλιάδες επιβάτες. Γνωρίζετε ότι έγινε μια τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα το πρωί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε εχθές το απόγευμα ε, σε, στο Συμβούλιο Μεταφορών. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω τα εξή Όλοι οι Υπουργοί Μεταφορών είναι υπέρ μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση στην κρίση. Οι εθνικές λύσεις ε, δεν ε, είναι επαρκείς να την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων που επηρεάζουν παγκοσμίω την κατάσταση αέρας κυκλοφορίας και το πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ των ε, Υπουργών Μεταφορών ήταν έντονο, είχαμε πολλές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, ε, όλοι ήταν έτοιμοι να αναλάβουν ευθύνη και να συνεργαστούν. Η ασφάλεια όμως έρχεται πρώτη. Είναι το σημαντικότερο δεν είναι δυνατόν ε, να κάνουμε κανένα σκόντο σε αυτό το θέμα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας ε, για τους επιβάτες μας. Επομένω, οι ε, Υπουργοί αποφάσισαν μια σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων και της και κυκλοφορίας. Άρχισε σήμερα το πρωί ε, γιατί σήμερα το πρωί η Eurocontrol ε, όρισε τρεις ζώνες ε, ανάλογα με την μόλυνση. Η πρώτη ζώνη αφορά τον κεντρικό πυρήνα των εκπομπών και σημαίνει πλήρη περιορισμό των πτήσεων όταν δεν υπάρχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια των αεροσκαβών. Δεύτερον, ζώνες ε, στις οποίες ε, θα γίνουν πτήσεις παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται η φεστιακή τέφρα ε, οι αποφάσεις βέβαια θα ληφθούν με συντονισμένο τρόπο μέσω των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και υπάρχει και μια ζώνη η οποία δεν ε, έχει καμία συγκέντρωση θεσιακής τέφρας και συνεπώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις πτήσεις ε, και βέβαια κάθε έξι ώρες ανατροφοδοτούνται οι πληροφορίες και διαβιβάζονται στις εθνικές αρχές. Περιμένουμε την ε, εφαρμογή ενός προγράμματος ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και βεβαίως των σχετικών δικτύων ε, και υπολογίζω βέβαια στην ε, υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ολόκληρο αυτό το πακέτο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού που ξεκίνησε πέρυσι. Γνωρίζετε και ο Υπουργό το ανέφερε μάλιστα ότι μια ομάδα δράσης, μια task force, μια ομάδα επιτρόπων οργάνωσε συζήτηση για το θέμα αυτό. Εχθές μίλησα με τους εκπροσώπους των ε, ε, αεροπορικών εταιριών και μας είπαν ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να εκτιμήσουν τις απώλειες, τις οικονομικές συνέπειες και ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης είναι να, ε, να ξαναγίνουν πτήσεις και δεν θα έπρεπε να πανικοβληθούμε με, με μέτρα κρατικών ενισχύσεων ή οτιδήποτε άλλο για την ενίσχυση του τομέα. Ένα σημαντικό ζήτημα βέβαια είναι τα δικαιώματα των επιβατών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την, το σεβασμό των δικαιωμάτων των επιβατών ε, γιατί όλοι συμφωνούν ότι οι κανόνες καλό είναι να υπάρχουν αλλά το ζήτημα είναι να ισχύουν και να εφαρμόζονται κάτι το οποίο βέβαια επαφίεται στα κράτη-μέλη. Εκείνα είναι αυτά που πρέπει να ε, προωθήσουν την εφαρμογή αυτή. Έχουν και εκείνα κάποιες ιδέες ε, για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων αυτών. Θα ήθελα τώρα να ε, σχολιάσω κάποιες ε, κατά τη γνώμη μου εσκεμμένες προσπάθειες να μπερδέψουν λίγο τα πράγματα ποιος έκανε τι, ποιος δεν έκανε τι και τι ακριβώς συνέβη. Είναι γεγονός ότι γίνονται εκλογές, ε, έρχονται εκλογές σε ορισμένες χώρες, αλλά μετά την έκρηξη του ηφαιστείου όλες οι αποφάσεις έγιναν βάση των μοντέλων λήψης αποφάσεων διαχείρισης των ζητημάτων αυτών. Και αποφασίστηκε η διακοπή αυτή. Υπάρχει λοιπόν ε, μία συνεργασία διακυβερνητική, αλλά ο εναέριος χώρος είναι κοινός. Ε, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή που αποφασίζει τους κανόνες των κρατών μελών, ούτε υπάρχουν περαιτέρω κανόνες όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των καταστάσεων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το μοντέλο αυτό. Συνεπώς, μπορούμε βέβαια να δούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε και αρχίσαμε ήδη να το συζητούμε από χθε αλλά το να λέει κανείς ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο απέτυχε πλήρως είναι εντελώς εσφαλμένο. Ήταν μια εντελώς ε, έκτακτη κατάσταση, κάτι το εντελώς απρόοπτο, ε, κάτι ε, το απρόσμενο, το γεγονός ότι εξαπλώθηκε τόσο πολύ η φεστιακή τέφρα είναι κάτι το οποίο δεν ε, ε, έχει συμβεί πολλές φορές, είναι εξαιρετικά σπάνιο, παγκοσμίω, δεν είναι κάτι σαν το χιόνι για παράδειγμα που είναι κάτι πιο σύνηθες. Το Σαββατοκύριακο φάνηκε ότι είναι μια πραγματικά πολύ εξαιρετική κατάσταση και ήδη κάναμε πολλές συζητήσεις για το πώς να προσεγγίσουμε την κατάσταση. Οι υπουργοί των μεταφορών είπαν κάποιοι θα έπρεπε να είχαν αμέσως παρέμβει. Μα κοιτάξτε, αυτό σε αυτό διαφωνούμε. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά είναι στα χέρια ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων ε, και εγώ και ο ε, Υπουργός Καρίδα επίσης μιλήσαμε με την Eurocontrol ε, την Κυριακή. Εγώ ήρθα σε επαφή με όλους τους ε, υπουργούς ε, των μεταφορών χωρών με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, για να το πω έτσι, για να μας πούν και εκείνοι ποια είναι η άποψή τους, τι θα έπρεπε να κάνουμε σε σχέση με την κατάσταση αυτή. Αλλά κοιτάξτε, δεν ήταν αυθαίρετες αποφάσεις αυτές που ελήφθησαν. Ειδικοί φορείς ε, αποφάσισαν, ε, συνεδρίασαν και έχουμε ήδη κάνει ε, πολλές συζητήσεις, ήδη από την Κυριακή. Μιλάμε για τη ζωή των ανθρώπων που διακυβεύεται εδώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και γι' αυτό ακριβώς τη Δευτέρα το πρωί έγινε και άτυπη συνεδρία του Συμβουλίου του Eurocontrol ε, και εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για το πνεύμα συνεργασίας που υπήρξε και σε σχέση βέβαια με το ε, μοντέλο αυτό των ε, τριών ζωνών τα γεγονότα λοιπόν δείχνουν ότι δεν μπορεί να υπάρχει μόνο εθνική προσέγγιση. Είναι παροχημένη μια τέτοιου είδους προσέγγιση καθαρά εθνική. Και συνεπώς θέλουμε να προωθήσουμε μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση για τέτοιου είδους ζητήματα και πρέπει βέβαια να εκτιμήσουμε και τις ε, συνέπειες ήταν, όλοι μας είπαν ότι το σημαντικότερο ήταν ε, να ξεκινήσουν και πάλι οι πτήσεις. Ε, όμως υπάρχει το θέμα, δηλαδή ότι έπρεπε να επιστρέψουν οι επιβάτες ε, στους προορισμούς τους. Και ότι αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα. Αυτό είναι κάτι που το συζητήσαμε. Ήταν το βασικό θέμα που συζητήσαμε χθες. Αυτά λοιπόν. Συνεργαζόμαστε και με το Συμβούλιο και με τη Eurocontrol ε, για να παρακολουθούμε την κατάσταση και αν χρειάζεται να λάβουμε νέες αποφάσεις. Αλλά για την ώρα το μοντέλο στο οποίο καταλήξαμε είναι αρκετά καλό για να ξεκινήσουν και πάλι οι περισσότερες πτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κάλλας. Και τώρα, έξω του ΕΛΚΕ, η κυρία Πόρτμαν Κόλ έχει το λόγο. Eh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις εξηγήσεις που έδωσαν και τα όσα είπαν όσον αφορά την κρίση στις ενέργειες μεταφορές στις τελευταίες ημέρες καταδείχθηκε σαφώς ότι όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προβλήματα όταν δεν υπάρχουν πτήσεις αλλά το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας όλοι οι πολίτες και η οικονομική ζωή πλήττονται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στην Ευρωβουλή να συζητηθεί αυτό το θέμα υπό τον χαρακτήρα κατεπήγοντο στην Ολομέλεια. Έχουν σταματήσει οι πτήσει, ε, οι επιχειρήσει, οι εταιρείε εναέριων μεταφορών ε, πλήττονται και υπάρχει αυτή η πτυχή στην οικονομική κρίση επιπλέον. Η ασφάλεια πρέπει να έχει πριτανεύοντα ρόλο, πρέπει να βρίσκεται πάνω-πάνω ω προτεραιότητα. Είναι φυσικό αυτό. Η ε, επιβάτες πρέπει με ασφάλεια να μεταφέρονται. Αλλά δεν είμαστε προετοιμασμένοι και εξοπλισμένοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση. Το κλείσιμο των αεροδρομίων και η πάυση των εναέριων μεταφορών ήταν μια πρώτη αντίδραση στο σύννεφο στάχτης. Όμως τα πρότυπα ε, στους ηλεκτρονικούς εγκεφάλους ε, δείχνουν ότι υπάρχει αυτό το σύννεφο, όμως έγιναν δοκιμαστικές πτήσεις και αρχίζει, μπορεί να αρχίσει το άνοιγμα των, του εναρίου χώρου αλλά με βάση πάντα ασφαλή δεδομένα και ασφαλή επιστημονικά τεκμήρια. Αυτά πρέπει τώρα να αξιολογηθούν και να μπορέσουν να διευρυνθούν. Πρέπει άμεσα να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Όμως οι ζώνες ασφάλειας, οι περιοχές αυτές πρέπει να μπορέσουν να ξανανοίξουν όταν θα είναι δυνατόν. Και υπάρχουν και διαθροτικά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Εδώ ε, υπάρχει η σε σχέση με το τον άνοιγμα του εναέριου χώρου. Όμω θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιδράσουμε γοργά. Οι εταιρείε εναέριων μεταφορών έχουν σημαντικές απώλειες που έχουν υποστεί. Όμως η υποστήριξη και περίθαλψη και φροντίδα των επιβατών είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Προστίθενται όλες αυτέ οι δαπάνε σε ύψο εκατομμυρίων ευρώ και πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει πρέπει γοργά να εξεταστεί και να αξιολογηθεί ποια, ποιο κόστος προκλήθηκε και πού είναι δυνατόν να υπάρξει ανακούφιση, αντιστάθμιση. Ένα παράδειγμα, όσον αφορά εταιρείε εναέριων μεταφορών, σε σχέση με την οδηγία περί δικαιωμάτων των ε, επιβατών ε, έδρασαν και πρέπει να δούμε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ε, θεομηνιών και τα λοιπά αν μπορέσει να υπάρξει δράση ο Επίτροπος Αλμούνια σε σχέση με αυτή την βοήθεια έχει δραστηριοποιηθεί. Θέλουμε όμως να πούμε ότι στόχος είναι οι εταιρείε να μπορέσουν να υποστηριχθούν μέσα σε ένα πλαίσιο όμως συντονισμού που θα ισχύει στην Ευρώπη και με βάση την πραγματική καταβολή αυτών των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ο κύριο Σούλτ, παρακαλώ σας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι αυτή η κρίση έχει και μια ανθρώπινη διάσταση για την οποία σίγουρα θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Δεν υπάρχουν λίγοι άνθρωποι, μυριάδες άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κολλήσει κάπου σε αεροδρόμια ελού και περιμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πρέπει να θυμηθούμε, να σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους ε, σήμερα το πρωί. Κάθε ένας από εμά είχε κάποια παρόμοια περίπτωση που έζησε, που βίωσε αυτό το τελευταίο διάστημα είμαστε ευρωβουλευτέ και έχουμε κάποια υποδομή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμεί ω ευρωβουλευτέ. Πάρα πολλοί όμω, μοιριάδε βρίσκονται, έχουν κολλήσει αλλού, δεν μπορούν να γυρίσουν στον χώρο εργασία του, δεν μπορούν τα παιδιά του να πάνε στο σχολείο, έχουν μείνει χωρί χρήματα, χωρί περίθαλψη, χωρί φροντίδα. Πρέπει να εκφράσουμε πραγματικά την, ε, ε, α το πω έτσι, αλληλεγγύη μα προ αυτού του ανθρώπου και να συναισθανθούμε τα προβλήματά του οι ε, επιχειρήσεις εναέριων μεταφορών είναι, λειτουργούν μέσα, μέσα σε ένα σύστημα ολόκληρο. Είναι συστημικά λοιπόν ε, θα έλεγα συγγενείς επιχειρήσεις. Όχι μόνο μεταφέρουν επιβάτες αλλά και αγαθά. Και είναι σαφές ότι οι απώλειές τους είναι πολύ σημαντικότερες από ότι σε σχέση με το πλήγμα της 11ης Σεπτεμβρίου του τρομοκρατικού πλήγματος στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν. Πρέπει να δούμε εδώ να υπάρχει ελαστική αντίδραση, ταχεία ανταπόκριση ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι εναέριες μεταφορές είναι τμήμα ενός δικτυωμένου πολύ ευρύτερου ε, συνόλου των, ε, στις διαθρώσεις, στη διάθρωση των ε, υποδομών και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τις ζημίες που προκλήθηκαν. Γι' αυτό η ιδέα που υπήρξε πριν από 20 χρόνια, η διεύρυνση των ευρωπαϊκών των ε, διαδικτύων, ιδιαίτερα η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου υποδομών σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο σιδηροδρόμων είναι κάτι πολύ σημαντικό σκέψη. Πρέπει τώρα να δώσουμε συνέχεια και να υλοποιήσουμε. Ο συνάδελφος Χαντράουι θα αναφερθεί σχετικά. Σήμερα δεν καταφέραμε να έχουμε διαλειτουργικότητα μεταξύ των τρένων των σιδηροδρόμων μεταξύ ε, των χωρών μας. Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να ταξιδεύει ένα γαλλικό τρένο υψηλής ταχύτητας μέχρι τη Βουδαπέστη, από τη Γαλλία μέχρι τη Βουδαπέστη ή να περνάμε εμεί από τη Γερμανία μέχρι την Ισπανία. Πρέπει λοιπόν εδώ να μην αντιδρούμε πυροσβεστικά και να αντιδρούμε μόνο στην αντιμετώπιση κάποιων αναγκών, αλλά να έχουμε ένα ευρύτερο συντονισμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δρούμε προ όφελο όλων. Η κυρία Μάισνερ, Γκεζίν Μάισνερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και κύριε Υπουργέ ε, από την Ισπανική Προεδρία. Είδαμε ότι η φύση είναι ισχυρότερη από όλη την τεχνολογία. Κατά κάποιο τρόπο εδώ οι άνθρωποι πήραμε ένα σοβαρό μάθημα από αυτή την κατάσταση. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε όμως επίσης ότι σε αυτή την περίπτωση είδαμε ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Εδώ και 20 χρόνια κάνουμε λόγο για την εσωτερική αγορά και για τις μεταφορές. Κάνουμε ε, λόγο για τον ενιαίο ε, ευρωπαϊκό ουρανό. Ίσως όμως με καλύτερο τρόπο θα έπρεπε να είχαμε συντονιστεί για να αντιδράσουμε σε σχέση με αυτό το ηφαίστειο. 20 χρόνια θέλουμε να υπάρξει, αυτός ο, να υπάρξει ο συντονισμένος ευρωπαϊκός ουρανός υπό το Ευρωκοντρόλ και δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Όπως και ο κύριος Σούλτς πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα με συντονισμένο τρόπο στις, ε, στους σιδηροδρόμους. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κράτηση για παράδειγμα απλά μέσω ε, σιδηροδρομικών ε, εταιριών ε, από τον βορρά στον νότο. Λείπουν λοιπόν εδώ αυτά τα στοιχεία και οι υποδομές. Πρέπει να πούμε ότι για τους πολίτες ήταν κάτι πραγματικά που δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Φυσικά ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση και δεν μπορούσε κανένας εθνικός Υπουργό να απελευθερώσει τον εναέριο χώρο όταν ε, υπήρχε το ε, πρόβλημα της ε, ανεπαρκούς ασφάλειας. Και έχουμε και το πρόβλημα της μη επαρκούς, ας το διασύνδεσης. Και έχουμε εδώ και τη δυσφορία των πολιτών και την οργή των πολιτών. Μπορεί να κατανοήσει κανείς και την θέση των, ενέριων, των εταιριών ενέριων μεταφορών που έχουν πληγεί και έχουν υποστεί ζημιές. Φυσικά υπάρχουν αυτέ οι ζημίες και είναι πολύ σημαντικό να γυρίσουν οι επιβάτες στα σπίτια τους. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους. Αλλά για τους επιβάτες στην Ευρώπη είναι σημαντικό να υπάρξουν δυνατότητες προσφορές ε, στις μεταφορές ε, για να μπορέσουν να επιστρέψουν. Πρέπει να υπάρξουν δηλαδή δυνατότητες ε, στις μεταφορές που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τι σημαίνει σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε συνέχεια και να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Στην κρίση που βρίσκεται και αντιμετωπίζει ο τομέας των μεταφορών ούτως ή άλλως, πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις εταιρείε εναέριων μεταφορών, να δώσουμε την δυνατότητα στους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματα ελευθερίας κυκλοφορίας και ε, Και ε, σε σχέση με τις ε, ε, αποζημιώσεις δεν είναι δυνατό να ζητηθεί να, από το ηφαίστειο να καταβάλει αποζημιώσεις. Η φύση δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη και να καταβάλει αυτές τις αποζημιώσεις αλλά προς το συμφέρον των πολιτών εμείς πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Γι' αυτό το βρίσκω πολύ καλό ότι δημιουργείται μια ειδική ομάδα δράσης Task Force υπό την αιγίδα του Προέδρου και με τη συμμετοχή των αρχών και του κυρίου Κάλλας θα δούμε και θα δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης για το μέλλον και πώς θα δράσουμε για να την αντιμετωπίσουμε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κυρία. Και εξ ονόματος τώρα των φιλελευθέρων και δημοκρατών που ο, ο, ο κύριος Κρέμα τώρα, εξ ονόματος των Πρασίνων και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Η κινητικότητα στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες ε, έχει αλλάξει με σημαντικό τρόπο. Δεν ήταν κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα, ούτε οι κλιματικές αλλαγές ή η ακριβή βενζίνη. Αίτιο ήταν αυτή τη φορά η ίδια η φύση. Το ηφαίστειο στην Ισλανδία έδειξε στην ανθρωπότητα για άλλη μια φορά ποια είναι η δύναμη της φύσης. Αυτό μας είναι μάθημα για το μέλλον. Δεν υπάρχει η υπερεξουσία, η μεγάλη αυτή ε, δύναμη των ανθρώπων που να επιβάλλονται στη φύση. Η φύση επιβάλλεται στους ανθρώπους. Επειδή η στάχτη αυτή μπορεί να σταματήσει τους κινητήρες ε, των ε, αεροπλάνων. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Eurocontrol με αίσθημα ευθύνη έδρασε και έθεσε την ασφάλεια των επιβατών ως ανώτατη προτεραιότητα. Εξ ονόματος των Πρασίνων θα ήθελα να ευχαριστήσω την Eurocontrol αλλά και την υποστήριξη των Υπουργών Μεταφορών και ιδιαίτερα όσον αφορά τον Γερμανό Γερμανό Υπουργό Μεταφορών, κ. Πέτα Ραμζάουερ. Θα ήθελα να πω ότι Πρέπει να υποστηριχθεί ακόμα και το Συνδικάτο των Πιλότων Cockpit που στην Γερμανία είναι, δείχνουν ε, αίσθημα ευθύνης και απορρίπτουν ε, προτάσεις ε, που μπορεί να μην είναι αξιόπιστες. Είτε θα είναι ο ενέργειο χώρος ασφαλής είτε δεν θα είναι ασφαλής. Και έτσι καταδικάζουν οι πράσινοι με κάθε οξύτητα την προσπάθεια των εταιριών να σημειώσουν κέρδη χωρίς να θέτουν την ασφάλεια των επιβατών σε πρώτο σημείο. Ζητούμε ο εναρίος χώρος στην Ευρώπη να απελευθερωθεί όταν οποιοδήποτε κίνδυνος θα μπορεί να αποκλειστεί. Ζητούνται όλοι οι πολιτικοί να είναι στεναροί και να μην υπαναχωρήσουν, να μην καμφθούν από την πίεση των εταιριών εναέριων μεταφορών. Πρέπει όμως να πούμε ότι ήταν οδυνηρό το έλλειμμα των ε, ελλείψεων που υπήρχαν τις τελευταίες ε, δεκαετίες που κάποιοι πίστευαν ότι μπορούσαν το σιδηρόδρομο να τον παραμελήσουν. Αυτή η πολιτική βασιζόταν οπωσδήποτε πλήρως ε, στις εναέριες μεταφορές. Παίρνουν 14 δις ετήσια οι εταιρείε εναέριων μεταφορών λόγω της μη εισπραξής ε, του φόρου επί της κυροζήνης. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πλήξει και τους σιδηροδρόμους ε, ταυτόχρονα. Όμως ένα μάθημα πρέπει να συναγάγουμε. Οι σιδηρόδρομοι δεν είναι μόνο το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, είναι το αναγκαίο μέσο για την διασφάλιση της κινητικότητας και το μέσο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να γίνει η προσπάθεια να επιστρέψουν στις, στα σπίτια τους οι επιβάτες. Ας είναι ένα μήνυμα συναγερμού η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία για το μέλλον των μεταφορών. Το μέλλον των μεταφορών θα το διασφαλίσουμε μόνο όταν δεν θα δρούμε με τρόπο πυροσβεστικό. Γι' αυτό ζητούνται από τα κράτη-μέλη να τεθούν προτεραιότητες στις μεταφορές με διαφορετικό τρόπο. Οι σιδηρόδρομοι δεν θα πρέπει μόνο με τα λόγια, αλλά και με χρηματοοικονομική υποστήριξη να τύχουν υποστήριξη για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρο, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών ο κύριος Βίτε παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη είναι η επιρροή του καιρού, των καιρικών συνθήκων και των κλιματικών συνθήκων ένα μικρό ηφαίστειο εξεράγει στην Ισλανδία, όμως ε, το σύνολο των εναέριων μεταφορών στην Ευρώπη έχει παραλύσει και αυτό εδώ και πολλές ημέρες. Είναι καλό ότι σήμερα υπάρχει έστω και εν μέρη α, νέα ανάκαμψη στις μεταφορές και έχουν ξεκινήσει κάποια δρομολόγια ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, συνθήκες ορατότητας που με, ορατότητας που με τις σημερινές ε, τωρινές ε, κλιματικές, κλιματικές συνθήκες μπορεί να πει κανείς ότι έχουν βελτιωθεί. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό όμως παραλύσει. Εδώ η υπέρπτυση για παράδειγμα μέσω των, ε, της εταιρείας ε, KLM ε, μέσω της Αλάσκας ή όταν είχαμε και προβλήματα με εκρήξεις ηφαιστείων στην Ινδονησία όμως αυτές οι πτήσεις πέρασαν πάνω από τη στάχτη ενός ηφαιστείου που μόλις είχε ξεκινήσει ε, η έκρηξή του. Δεν μπορεί να συγκριθεί η κατάσταση εκείνων των υπερπτήσεων ε, ηφαιστείων με την κατάσταση που έχει προκληθεί στην Ευρώπη με το, την έκρηξη του ηφαιστείου της Ισλανδίας που έχει ε, καλύψει τους ουρανούς της Ευρώπης με στάχτη. Και έτσι λοιπόν εξαρτάται η απόφαση αν θα απελευθερωθεί ο εναέριος χώρος ανάλογα και με το ύψος στο οποίο διεξάγεται μια πτήση. Λόγω του ότι η στάχτη από το ηφαίστειο αυτό της Ισλανδίας ε, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην οικονομία της ε, Ευρώπης ε, και στις εναέριες μεταφορές που έχουν πληγεί. Οι μεγάλες εταιρείες ίσως μπορούν να τα καταφέρουν, όμως πρόκειται για πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση σε σχέση με τη στάχτη του ηφαιστείου και να δούμε αν θα υπάρξει άνοιγμα αεροδρομίων και εναερίων ζωνών. Θα πρέπει να πούμε ότι οι ασφαλείς μεταφορές ε, μπορούν να λειτουργήσουν όταν σταθμίζουμε τα συμφέροντα της ασφάλειας και της οικονομίας σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και στη συνέχεια ο Λόταρ Μπίσκι από την Ενωτική Αριστερά. Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση της ε, υπηρεσίας για την ασφάλεια των εναέριων μεταφορών η ασφάλεια των επιβατών να είναι η πρώτη προτεραιότητα και να μην διακυβευτεί ήταν σωστή υπόθεση. Ακόμα και αν αυτό συνεπαγόταν το κλείσιμο του εναέριου χώρου για πολλέ ημέρε. Ακόμα και αν αυτό σήμαινε θυσίε οικονομικέ και απώλειε για τι εταιρείε εναέριων μεταφορών. Εγώ νομίζω ότι είναι ανεύθυνο οι εταιρείε εναέριων μεταφορών να αφήσουν του πιλότου του να πετούν σήμερα με, δικό του κίνδυνο, με δική του ευθύνη. Τι σημαίνει εδώ με δική του ευθύνη. Το χαιρετίζω ότι εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυση των εταιριών εκείνων που χωρί βοήθεια θα βρισκόντουσαν σε πολύ δυσχερή κατάσταση. Θα συζητήσουμε και για την κατάσταση στην απασχόληση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να αποφευθεί μια περαιτέρω οικονομική επιδείνωση των πραγμάτων, αυτό θα είναι σωστό αντισταθμίζοντας τα πράγματα σε σχέση με την έγκριση επιδοτήσεων ή ενισχύσεων θα πρέπει δεσμευτικά να συμφωνηθεί ότι οι εταιρείε εναέριων μεταφορών δεν θα προβούν σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού τους ε, και δεν θα προβούν σε μείωση και των μισθών των εργαζομένων τους. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό δεν θα ε, στερηθεί οι μέρες ε, από τις απολαβές του όσον αφορά τις διακοπές του, τις πληρωμένες διακοπές του και έτσι σε σχέση με δυσκολίες που είχαν κάποιοι να παρουσιαστούν στο χώρο εργασίας τους επειδή είχαν κολλήσει σε αεροδρόμια να μην υποστούν αυτές τις θυσίες. Πρέπει εδώ να μπορέσει να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή επιτήρηση του εναριού χώρου προς όφελος της ασφάλειας. Ρητά και κατηγορηματικά αυτή η εποπτεία θα πρέπει να στοχεύει κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ. Υπενθυμίζω εδώ τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ των τραπεζών που α το πω έτσι κέρδισαν, αποκόμισαν ήταν κέρδη από την κρίση, όμως δεν δραστηριοποιήθηκαν με κοινωνικό πνεύμα και κοινωνική στοχοθέτηση. Ο ανταγωνισμός και η κερδοφορία δεν μπορούν να έχουν την ανώτατη προτεραιότητα και έναντι μάλιστα της ασφάλειας των ίδιων των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο συμπρόεδρος κύριος Περώνη. Ευχαριστώ. Κατ' εμέ η κατάσταση που δημιουργήθηκε από το ηφαίστειο καθυστέρησε να ε, αντιμετωπιστεί και η πρώτη συνεδρίαση επίσημη έγινε τη Δευτέρα. Η έκρηξη του ηφαιστείου και η ηφαιστειακή τέφρα ξεκίνησε να υπάρχει την Πέμπτη το πρωί. Πέντε μέρες για να ε, ληφθεί μία αποτελεσματική απόφαση. Ίσως ελήφθησαν ε, αποτελε... υπερβολικά μέτρα. Κατά πρώτο λόγο η ασφάλεια. Γιατί να απαγορεύσουμε όμως τις πτήσεις στο Βέλγιο όταν το νέφος είναι στην Ορβηγία. Γιατί να απογορευτεί η πτήση των μονοκινητών κινητήριων αεροπλάνων στα 450 μέτρα όταν ε, η τέφρα ήταν άνω των 8.000 μέτρων εφαρμόστηκε ίσως ε, ο κανόνας ε, που γνωρίζουμε εμείς οι πιλότοι εδώ και χρόνια είναι ο κανόνας που λέει ότι ο πιλότος πρέπει να είναι στο μπαρ και το αεροπλάνο πρέπει να βρίσκεται στο υπόστεγο. Αλλά δεν είναι έτσι η κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν για να διασφαλίσουμε την ε, ασφαλή μετακίνηση των επιβατών και των πιλότων και των πληρωμάτων, ναι μεν θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, αλλά επαναλαμβάνω τα μέτρα ήταν πάρα πολύ καθυστερημένα σε σχέση με την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν για το μέλλον να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες ασφάλειας καταρχάς καθώς επίσης και τις ανάγκες οι οποίες ε, σε συνδυασμό με την ασφάλεια δεν θα κάνουν αδιακρίτως απαγόρευση των πτήσεων, αλλά θα λαμβάνονται μέτρα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη στην πραγματική κατάσταση, όχι τη στατιστική κατάσταση. Διότι θα πρέπει να επιτρέπεται σε ένα ζωτικό, νευραλγικό ε, τομέα για την οικονομία να μπορεί να λειτουργήσει. Διότι οι οικονομικέ επιπτώσει δεν θα είναι μόνο στον αέριο χώρο και στι αεροπορικέ εταιρείε και το τομέα του τουρισμού, αλλά για όλη την οικονομία. Το διαπιστώσαμε αυτό όταν είχαμε και την 11η ε, ε, Σεπτεμβρίου και την πτώση των δίδυμων πύργων. Σας καλώ λοιπόν να δράσετε κατεπηγόντως, σοβαρά και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος ε, των μη εγγεγραμμένων. Η κυρία Αγγέλικα Βέρτμαν παρακαλώ, έχει τον λόγο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα ο κίνδυνος μια, ένα αεροπλάνο με επιβάτες, γεμάτο επιβάτες να πάθει μια βλάβη στους κινητήρες και να ε, πέσει στο έδαφος, να καταπέσει είναι τεράστιος. Υπενθυμίζω ότι υπήρξε υπέπτυση αεροπλάνου στο παρελθόν πάνω από ένα τέτοιο ε, ηφαίστειο που είχε εκραγεί και το 1989 ένα αεροπλάνο του, της KLM πέταξε πάνω από ένα ηφαίστειο που είχε μόλις ε, εκραγεί. Οι ανθρώπινες ζωές ε, δεν ε, μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα. Χαιρετίζω την απόφαση να ε, κλείσει ο ενέριος χώρος και έτσι να αφαιρεθεί από τους πιλότους η ευθύνη, η ιδία ευθύνη να κρίνουν κατηδίαν. Οι πραγματικές αναλύσεις και αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν σε κάποια καθοριστικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση της KLM υπήρχαν τέτοια σωματίδια στάχτης αλλά δεν ήταν ορατά. Ε, η φύση δείχνει ότι ακόμα και σε μια φάση παγκοσμιοποίησης ε, η ε, φύση έχει το πάνω χέρι. Ωστόσο η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανώτερη από την αξία των οικονομικών αγαθών. Γι' αυτό γνωρίζω, έχοντας υπόψη αυτά τα προηγούμενα συμβάντα ζητούμε να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στην αντιμετώπιση της κατάστασης τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα οι άλλοι αγορητές. Ο κύριος Ματίο Γκρός, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Αυτή η απαγόρευση ενεργείων μεταφορών οδηγεί σε αυτή την ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια σε εναέριες μεταφορές που έχει γίνει και αρκετές φορές στην Ευρωβουλή και που έχουμε καταδείξει ότι εμείς στην Ευρωβουλή και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλαμε και μπορέσαμε να δραστηριοποιηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν το επιθυμούσαν και το θέλουν τα κράτη-μέλη. Και αυτή τη συζήτηση δεν την έχουμε κάνει μόνο για τις ενέργειε μεταφορές αλλά και για του σιδηροδρόμους. Γι' αυτό πρέπει οι ερωτήσεις αυτές με θετικό τρόπο να μπορέσουν να απαντηθούν. Από τις ε, υπηρεσίες ε, για την ε, πολιτική αεροπορία και τον έλεγχο των εναέριων μεταφορών πιστεύω ότι τα πράγματα λειτουργήσαν καλά. Σήμερα η πρώτη προτεραιότητα είναι, πιστεύω εγώ, η ασφάλεια των επιβατών και όχι τόσο η οικονομική πτυχή, η κερδοφορία των εναέριων μεταφορών, παρότι και αυτό το σημείο δεν πρέπει να το αμελήσουμε. Στο μέλλον η πρώτον η Eurocontrol και δεύτερον οι εθνικές υπηρεσίες για την ασφάλεια των εναίριων μεταφορών πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις και όχι κάποιοι άλλοι και γι' αυτό να λαμβάνονται υπόψη οι απόψει των επαϊόντων. Οτιδήποτε άλλο είναι πολύ επικίνδυνο. Φυσικά υπό οικονομικό πρίσμα η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε μετά την έκρηξη του ηφαιστείου αυτού είναι ένα περαιτέρω οικονομικό πλήγμα το οποίο υφίστανται οι εταιρείε εναέριων μεταφορών. Και μετά το τρομοκρατικό πλήγμα της 11 η Σεπτεμβρίου και μετά την οικονομική κρίση που έπληξε παγκόσμια τόσες χώρες αλλά ιδιαίτερα και την Ευρώπη και βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες απώλειες. Ναι, να δοθεί βοήθεια, αλλά όχι μόνο σε κρατικό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο. Οι επιβάτες και έχουμε συζητήσει για αυτούς τόσες φορές στο παρελθόν στην Ολομέλεια της Βουλής, οι επιβάτες είναι εκείνοι οι άνθρωποι που πρέπει να βοηθηθούν, να μπορέσουν υπό το πλαίσιο του κειμένου δικαίου να τύχουν του, της μέγιστης βοήθειας ε, και έτσι να αντιμετωπιστούν οι επιβάτες με τέτοιο τρόπο από τις εταιρείε εναέριων μεταφορών ώστε να είναι σεβαστά τα δικαιώματά τους. Ε. Για το μέλλον για μας είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουράνιος χώρος, ε, εναέριος χώρος. Και πρόεδρε, αυτό το θέμα εδώ στην Ευρωβουλή πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι σημαντικό αυτό αυτούς τους επιβάτες που έχουν κολλήσει στα αεροδρόμια και στο εξωτερικό να τους ε, φέρουμε πίσω στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Ε, και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών έχει ένα ελάχιστο επίπεδο που προβλέπει για την ε, βοήθεια και την παροχή υπηρεσιών και φροντίδας σε αυτούς τους επιβάτες. Δημιουργήθηκε όμως ένα χάος στην Ευρώπη με αυτή την κατάσταση. Είμαι υπέρ του να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό σενάριο το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει ώστε να μπορέσουν να γνωρίζουν οι επιβάτες πώς θα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις στο μέλλον και πώς θα δραστηριοποιούμαστε ώστε να μπορούμε να τους βοηθούμε και να τους παράσχουμε την αναγκαία φροντίδα. Θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία task force, μία ειδική ε, μονάδα που θα δημιουργηθεί ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν αυτοί οι επιβάτες ε, στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους τους. Όμως κάποιοι επιβάτες που πρέπει ε, μεγάλες πτήσεις, μεγάλες αποστάσεις να καλύψουν, ίσως θα χρειαστεί ακόμα περισσότερο διάστημα να περιμένουν. Και τι θα γίνει σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση. Όλα αυτά απαιτούν περισσότερο ευρωπαϊκό συντονισμό. Επισημάθηκε ότι ο ευρωπαϊκός ενιαίος εναέριος χώρος θα μπορούσε να βοηθούσε αν είχε επιτευχθεί. Όμως δεν έχει άμεσες αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφασίσει για τον εναέριο χώρο χώρο μελών, ούτε η Eurocontrol. Γι' αυτό ο συντονισμός έχει τεράστια σημασία. Και χθε το βράδυ και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πρώτη φορά η δημιουργήθηκε, προτάθηκε ένα μαθηματικό πρότυπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το χάος αυτό ε, τα μικρότερα σωματίδια, τα ελάχιστα αυτά σωματίδια χρησιμοποιήθηκαν ως αφορμή για να κλείσει ο ενέριος χώρος. Στις ΗΠΑ οι Αμερικανοί αξιολογούν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Δημιουργούν αεροδιαδρόμους και με αυτόν τον τρόπο μεριμνούν ώστε να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί αυτό το πρότυπο και να δούμε τι μπορεί να γίνει από πλευράς, μα ε, μας στην Ευρώπη. Επίσης ε, να δούμε σε σχέση με την, τις αποζημιώσεις χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν θα πρέπει όμως να φανταστούμε ότι όλες οι ζημιές μπορούν να αποζημιωθούν και να καλυφθούν. Κάτι τέτοιο θα πήγαινε μακριά. Ο κύριος Στέρξ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ καταρχήν θα ήθελα πρώτα να στραφώ στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και να του πω το εξή. Και αυτό δεν απευθύνεται σε εσά προσωπικά, κύριε ε, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αλλά πρόκειται για το Συμβούλιο, για εσά ω Προεδρία και για την επόμενη Προεδρία. Πώ είναι δυνατόν να μην τα καταφέρνουμε ω Ευρωπαίοι. Πάντα αποτυγχάνουμε στο Συμβούλιο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο προσπαθούν να ασκήσουν την επιρροή του. Όμω στο τέλο τέλο το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο ε, στυλώνει τα πόδια και δεν ε, προχωρούμε. Ένα από τα μαθήματα που μπορούμε να συναγάγουμε από την κρίση είναι αυτό. Ο κύριο συνάδελφο ε, Χαντράου είπε ότι ο συντονισμό θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει καλύτερα. Όχι μόνο όσον αφορά τον χώρο, αλλά και ο συντονισμό μεταξύ των, ευρωπαϊκών, των ε, κρατικών αρχών για την ε, ασφάλεια των ε, μεταφορών, των εναέριων μεταφορών, θα έπρεπε ο συντονισμός αυτός να λειτουργήσει καλύτερα. Θα έπρεπε λοιπόν το Συμβούλιο να μπορέσει να διευκολύνει τα πράγματα. Ένα επιπλέον στοιχείο, οικονομικές πληροφορίες. Σε σχέση με ένα κέντρο στο Λονδίνο που θα μπορούσε να αποφασίζει αυτά τα θέματα με την Eurocontrol. Είναι θεμητό να θέλουμε να να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πρότυπο, να, συγκλίνουν, να συγκλίνουν τα διαφορετικά πρότυπα που έχουμε και να καταλήξουμε σε μια κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Διότι ε, τα ηφαίστεια δεν είναι κάτι το καινούριο. Εδώ και πολλά χρόνια, ε, επί δέκα χρόνια ε, βρισκόταν υποδιαρκή έκρηξη αυτό το ηφαίστειο. Πρέπει λοιπόν τα δικαιώματα των επιβατών να διασφαλιστούν και η κρατική ενίσχυση πρέπει μέσα σε, στα εύνομα πλαίσια να διαμορφωθεί. Κυρία Ντυρόμπα. Ευχαριστώ πολύ. Παρά το γεγονός ότι Χιλιάδε άτομα βρίσκονται σήμερα σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά μα ε, επαναφέρει στην τάξη η φεστιακή έκρηξη. Πρέπει να δούμε την κατάσταση όχι μόνο στι μεταφορέ, ε, αλλά και την εξάρτηση από τι ε, εναέριες μεταφορέ που έχει αντικαταστήσει του υπόλοιπου τρόπου μεταφορών. Κανένα δεν μπορεί να πει πότε θα σταματήσει αυτή η έκρηση και πώ το νέφος θα μετακινηθεί κατά τι επόμενε εβδομάδε και κατά του επόμενου μήνε. Γι' αυτό Υποστηρίζω και το Συμβούλιο και την Επιτροπή ε, ότι πρέπει να διατηρήσουμε την αρχή της πρόληψης και της ασφάλειας και πρέπει να δούμε τι συμβαίνει για παράδειγμα και με τον φαρμακευτικό τομέα γιατί πολλές φορές ε, εν ονόματι της πρόληψης ε, πιέσαμε τα πράγματα προς μια συγκεκριμένη κατέσταση. Σήμερα ένας άλλος τομέας καταγγέλει αυτή την πρόληψη των κρατών ή του Συμβουλίου. Νομίζω ότι η ασφάλεια είναι το σημαντικότερο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Και αυτό που επίσης δείχνει η κρίση αυτή είναι η σημασία του σιδηροδρομικού τομέα. Ε, δείχνει ακριβώς ε, πόσο θα έπρεπε να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς του σιδηροδρομικού τομέα στις μεταφορές. Δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα τρένα και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της Λευκής Βίβλου που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή ε, η Επιτροπή. Η αποζημίωση, ο πατρισμό των επιβατών είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να δούμε και στη συνέχεια τι θα κάνουμε πολύ στοχευμένα με τις ε, αεροπορικές εταιρείε στη συνέχεια. Πρέπει να υποστηρίξουμε πολύ περισσότερο την τηλεδιάσκεψη είναι κάτι το ε, δευτερογενές μεν, ε, αλλά σε γενικές γραμμές μας χρησιμεύσε και αυτό και μπορεί και να μας βοηθήσει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις ε, εναέριες μεταφορές. Ε, ο πρόεδρος το ανέφερε προηγουμένως, ίσως και το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να δει την, ε, να αναθεωρήσει την οργάνωσή, της, την οργάνωσή του. Για ποιο λόγο να μην δουλεύουμε πέντε, πέντε μέρες την εβδομάδα αντί για τρεις, για να μπορέσουμε να μην εξαρτώμεθα τόσο πολύ από τις εναέριες μεταφορές που φαίνεται είναι πολύ ευάλωτες και μας ε, σε πράγματα τα οποία δεν είχαμε, αντιμε... δεν είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και δεν έχουμε πείρα να τα αντιμετωπίσουμε. Η Λευκή Βίβλος λοιπόν για το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά πρέπει και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξουμε και άλλου τρόπου μεταφορών ε, και αυτό αναφέρεται και στον τρόπο εργασία των δικών μα. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λυπούμε για το γεγονός ε, ότι από ό,τι φαίνεται πολλοί από τους συναδέλφους πριν λάβουν το λόγο δεν ε, ζήτησαν τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Άνθρωπου, ανθρώπους που έχουν περάσει ώρες πτήσης ε, στα πιλοτήρια. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πολιτική συζήτηση και έχω την εντύπωση ότι ρίχνουμε τι ευθύνε στο, Συμβούλιο για την έγκριξη του ηφαιστείου. Δεν μπορούμε να επιρρύπτουμε ευθύνε για μια έγκριξη ευθυσίου σε κανόνα. Η απόφαση της Eurocontrol θεωρώ ότι ήταν ευεβιασμένη και το δηλώνω αυτό διότι ουσιαστικά ρίχνουμε όλα τα ε, πράγματα στο ίδιο σακούλι. Δεν λαμβάνουμε υπόψη την ποικιλομορφία της κατάστασης. Εγώ είμαι υπέρ μια ε, συνειδητή εποπτείας. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να προκύψει από όλη αυτή τη συζήτηση. Αλλά θεωρώ ότι οι αποφάσει οι οποίε ελήφθησαν θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν διαφορετικές. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Ανά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή και να συμπάσχουμε με όλους όσους ήταν ή είναι θύματα της κατάστασης αυτής. Επίσης πρέπει να συμπάχουμε και με τους μισθωτούς των εργαζομένων των αεροπορικών εταιριών που προσπάθησαν με τον τρόπο τους να υποστηρίξουν επιβάτες. Δεν συμφωνούμε με αυτούς που, που κρίνουν αλλά προτείνουν ε, λίγα πράγματα το να λέμε εδώ ότι η ασφάλεια πρέπει να ε, επιβεβαιωθεί ως προτεραιότητα. Πρέπει ε, να ξέρουμε ότι καλύτερα είναι να υπάρχουν άνθρωποι απογοητευμένοι και ταλαιπωρημένοι από, ε, από νεκρούς είναι πολύ σημαντικό ε, να είμαστε ενωμένοι. Ενδεχομένως αυτό θα μας είχε δώσει τη δυνατότητα να εξηγήσουμε περισσότερο ε, στους ανθρώπους που ζητούν πληροφορίες για την κατάσταση αυτή. Οι υπηρεσίες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να εξελιχθούν σε ένα επιστημονικό συμβούλιο που θα μπορούσε να υποστηρίξει σημαντικές αποφάσεις στο μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, πρέπει να εργαστούμε ακόμη περισσότερο για τη συμπληρωματική συμπληρωματικότητα των τρόπων μεταφορών ε, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη συνοχή των ε, μέσων μας ε, για να μην υπάρχουν πλέον υποψίες που ενδεχομένως να υφίστανται ακόμη και πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια ερευνητική επιτροπή του θέματος αυτού από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Άννα Ρόσπαχ. Για 1,5 λεπτό. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Εδώ τίθενται κάποια πιεστικότατα ερωτήματα. Πρώτον, οι ενέργειες μεταφορές έχουν παραλύσει και δεν είναι ανταγωνιστικές. Αλλά αυτό ισχύει και για τις αμερικανικές και για τις ασιατικές εταιρείες που δεν μπορούν να προσγειωθούν στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι απώλειες κατανέμονται σε όλους. Τώρα, τίθεται το θέμα της αντιστάθμισης ή των αποζημιώσεων για τις εταιρείες ενέργειων μεταφορών. Περί αυτού θα πρόκειται τις επόμενες ημέρες. Χαίρομαι τώρα ότι υπάρχει προσέγγιση σε σχέση με τις ε, διαφορετικές ε, ζώνες. Ε, στην Financial Times υπάρχει, υπάρχουν επικρίσεις σε σχέση με τους πολιτικούς που λόγω φόβου λέει έκλεισαν τον ενέργειο χώρο και θα πρέπει λέει να αποφασίζουν οι ίδιες οι εταιρείες ενέργειων μεταφορών. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απορρίψει μια τέτοια προσέγγιση. Θα ήταν ολέθριο αν επιτρέπαμε κάτι τέτοιο ως προσέγγιση και αν μόνο για λόγους κερδοφορίας οι εταιρείες ενέργειων μεταφορών συνέχιζαν τις πτήσεις τους και αυτό μάλιστα με κίνδυνο των επιβατών. Τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εξελίξεις, να σημειωθεί πρόοδος, να αναπτυχθούν νέοι κινητήρες για τα αεροπλάνα που δεν θα είναι τόσο ευπαθείς. Αλλά όμως οι εναέριες μεταφορές συνολικά είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, όχι μόνο εναντί πληγμάτων από τους ε, ε, χτυπημάτων από τους τρομοκράτες, αλλά και λόγω φυσικών καταστροφών και θεομηνιών. Χρειαζόμαστε άλλες εναλλακτικές δυνατότητες. Και επιτέλους ε, τα τρένα υψηλής ταχύτητας να τα εκμεταλλευτούμε και να διευρύνουμε τα δίκτυά τους περισσότερο και να υπάρξει και διαδικτύωση μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, των μεγάλων πόλεων και να μπορέσουμε έτσι με ασφάλεια να ανταγωνιζόμαστε τις εναέριες μεταφορές με τους σιδηροδρόμους. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά τώρα η κυρία Hübner. παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε ε, Επίτροπε, Σήμερα γνωρίζουμε καλύτερα από ότι πριν από κάποιες μέρες ε, ότι υπάρχει τεράστιο κόστος. Ε, έχουμε και το θέμα το οποίο ξεπερνά τις απώλειες ε, των ενάριων μεταφορών. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτό το νέο πλήγμα έπληξε την ήδη πάρα πολύ ευάλωτη ευρωπαϊκή οικονομία βλέποντας το θέμα των, της οικονομικής αντιστάθμισης σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις που θα πρέπει να προσφέρεται στις εναέριες μεταφορές. Έχουμε και ένα προηγούμενο από πλευρά των Αμερικανών μετά το τρομοκρατικό πλήγμα της 11 Η Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν δράση από πλευρά της Ευρώπης. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γνωρίζουμε το αναμενόμενο αυτό βάρος, την αναμενόμενη επιβάρηση όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας και τα δημοσιονομικά μας που ήδη έχουν πιεστεί πάρα πολύ και πιέζονται σε σχέση με την βοήθεια μέσω αυτών των κονδυλίων από τον προπολογισμό μα. αυτό είναι η μόνη λύση ή υπάρχουν και άλλε εναλλακτικέ δυνατότητε. Δεύτερη ερώτηση αφορά το δυναμικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων. Ακούμε ότι τι πρώτε ημέρε δεν υπήρξε συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών σε μια κατάσταση που κάλυπτε πάνω από 80% του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία αλλά και να υπάρχει και συντονισμός. Αυτό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στην ε, υιοθέτηση καλύτερων ε, λύσεων. Θα πρέπει λοιπόν σε σχέση με μια νέα αντιμετώπιση και ε, διαχείριση κρίσεων να δούμε ότι αυτά μπορούν να συμβούν, αυτά τα πλήγματα μπορούν να συμβούν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Γι' αυτό ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το έναυσμα αυτή τη καταστροφή ώστε να διευρυνθεί το δυναμικό και η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδρά αποτελεσματική. αποτελεσματικά. Θα βοηθήσουμε εμείς εσάς για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ο κύριος Χάνες Βόμποντα παρακαλώ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Τι τελευταίε ημέρε. Τι εναλλακτικέ λύσει για τι εναερίε μεταφορέ στην Ευρώπη τι είδαμε και τι ζήσαμε και τι βιώσαμε και σε σχέση με μια διαδρομή από το Βελιγράδι στη Βιέννη και από τη Βιέννη στο Στρασβούργο. Και όσον αφορά το οδικό δίκτυο είναι σχετικά καλά ανεπτυγμένο και στι συνοριακέ περιοχέ. Όμω ε, ο σιδηρόδρομο εξακολουθεί να είναι σε μια δεινή κατάσταση και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Τι γίνεται σε σχέση με τα σχέδια του προγράμματος, του σχεδίου Delors. Αν είχαν υλοποιηθεί αυτά θα είχαμε περισσότερα τρένα υψηλής ταχύτητας, αποτελεσματικούς σιδηροδρόμους μετά από λίγες ώρες δεν μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει τις τουαλέτες ε, στα βαγόνια στο σιδηρόδρομο γιατί επί ώρες ε, βρισκόντουσαν ε, υπερβολικά πολλοί επιβάτες σε αυτά τα τρένα και δεν επαρκούσαν οι τουαλέτες. Παρακαλώ λοιπόν τον Επίτροπο να δοθεί μια νέα όθηση στον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων με περισσότερα τρένα υψηλής κατάστα... ταχύτητας. Χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο δυναμικό για τους σιδηροδρόμους. Και αυτό όχι μόνο σε σχέση με αυτή την καταστροφή με το ηφαίστειο αλλά και το χειμώνα ακόμα. Βλέπουμε ότι δεν επαρκεί η παροχή υπηρεσιών από πλευρά των σιδηροδρόμων για του πολίτε μα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, συνάδελφε. Για 1,5 λεπτό η κυρία Βιλμπάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Γκαρίντο και τον κύριο Κάλλας για τις εξηγήσεις και για τις προσπάθειές τους. Συμφωνώ μαζί σας ότι η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια, ότι πρόκειται για μια πολύπλοκη κρίση, αλλά ότι καθυστερήσαμε με την επικοινωνία, διότι ε, η πρώτη ανακοίνωση ε, προέκυψε πέντε, πέντε μέρες μετά από την έκρηξη. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά που περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από εμά, οι αποφάσεις πρέπει να είναι απλές, ε, και να μπορούν να εφαρμοστούν και να έχουν και επιπτώσεις οποίες θα μπορούν να τις αντιληφθούν όλοι. Όλοι όσοι συνεισφέρουν, όλοι όσοι θα πρέπει να καταβάλουν το τίμωμα για αυτή την κρίση θα πρέπει να τους εγγυηθούν τρία πράγματα. Μεγαλύτερη διαφάνεια για τις αποφάσεις για το κλείσιμο των αεροδρομίων και για την εξέλιξη της κατάστασης διότι ανακοινώθηκαν καθυστερημένα όλες αυτές οι ανακοινώσεις τις πρώτες ώρες της κρίσης και αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν τα προβλήματα και μάλιστα χωρίς λόγο στο αεροδρόμιο και δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα προβλήματα για πολλούς επιβάτες προκειμένου να ε, βρουν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης. Τώρα που καθορίστηκαν αυτές οι τρεις περιοχές θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι αυτές και πώς ακριβώς θα εξελιχθούν. Όσον αφορά τώρα στα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για, τα δικαιώματα των, ε, για να καταβάλουν το αντίτιμο για τα δικαιώματα των επιβατών και σε τι προθεσμίες θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Συμφωνώ επίση και με τον Επίτροπο Κάλλα ε, στο ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία συνέχεια τη διαδικασία και να δούμε τι θα κάνουν οι αεροπορικέ εταιρείε για να αντιμετωπίσουν τι αιτήσει αποζημίωση. Και τέλο, για τι κρατικέ ενισχύσει προ αεροπορικέ εταιρείε. Θα ήθελα να καθορίσουμε σαφώ ποιε θα είναι αυτέ οι βοήθειε, με τι κριτήρια θα δοθούν και να συνεχίσουμε να ελέγχουμε και τις πιθανές επιπτώσεις τις οποίες θα μπορεί να έχει αυτή η κρίση για τους εργαζομένους των αεροπερικών εταιριών. Θα πρέπει επίσης να αυξήσουμε τα μέτρα ασφαλείας ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να μην μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να μπορέσουν να, κάνουν, ε, ε, να λάβουν υπερβολικά μέτρα κατά των εργαζομένων. Η κρίση μας έχει δημιουργήσει μια κατάσταση ανασφάλειας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριος Μπράντμπουν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως είπαμε ήδη, κανένας δεν θα μπορούσε να προβλέψει τα όσα συνέβησαν στην Ισλανδία και οι αεροπορικέ εταιρείε βρέθηκαν ενώπιον απρόσμενων καταστάσεων και λόγω της έκρηξη του ηφαιστείου φυσικά και λόγω της οικονομικής κατάστασης ελήφθη εν ώψη αυτή τη κατάσταση ένα ακραίο μέτρο κλεισίματο όλων των αεροδρομίων χωρί επιστημονικέ γνωμοδοτήσει και από τα όσα λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι οι διαταραχέ ήταν ελάχιστε και δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα. Οι αεροπορικέ εταιρείε ε, δημιούργησαν περαιτέρω απογοήτευση διότι είχαμε κακή διαχείριση τη κρίσεω. Το να δίνονται μέτρα και νέε ανακοινώσει κάθε έξι ώρες σημαίνει ότι ούτε οι ίδιοι οι επιβάτες ήξεραν τι πρέπει να κάνουν και πώ μπορούσαν να προγραμματίσουν και οι αεροπορικέ εταιρείε ε, βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση. Παρά το γεγονό ότι υπάρχει μεγάλη τεχνολογία, υπάρχουν δορυφόροι, συστήματα, τεχνικά ε, μέσα, ε, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου τελικά βγάζαμε το δάχτυλό μα έξω από το παράθυρο για να δούμε αν φυσάει αέρα. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση θα πρέπει να μας ηχεί όλους. Μακροπρόθεσμες προγνώσεις ε, χρειαζόμαστε και κατάλληλα μέτρα μετεωρολογικά. Δύο, ε, λεπτά για την κυρία Κριστίν Τεβεράκ. Merci, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω ότι η πρόληψη την οποία ανέφεραν οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κλείνοντας τον εναέριο χώρο με στοχευμένο και στοχευμένα και προσωρινά ήταν ε, συνετή απόφαση γιατί η ασφάλεια των πολιτών ε, είναι ανώτερη από οτιδήποτε άλλο και το γεγονός ότι κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείε λένε ότι μπορούν να ανοίξει αμέσως πλήρως ο εναέριος χώρος ε, είναι κάτι το απαράδεκτο κύριος Ενάν προηγουμένω μίλησε για τη συμπληρωματικότητα των ε, μέσων ε, μεταφοράς ε, και κυρίως για το τρένο. Πραγματικά θλίβομαι που η εναέρια παράλυση ε, μερικές φορές, για παράδειγμα στη Γαλλία, ε, είχε ως αποτέλεσμα ε, την υποτίμηση της, του τρένου με ανεύθυνο τρόπο. Ε, η αναστάτωση βέβαια είχε, ως, ε, είχε, είχε προκύψει από την ανάγκη της ασφάλειας, της ασφάλειας των επιβατών και γι' αυτό προτείνω μεταξύ των κριτηρίων ε, για το άνοιγμα του εναερίου χώρου να είναι η αποζημίωση που προτείνουν οι αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση ακύρωση της πτή, ακύρωσης πτήσης γιατί υπάρχει και η ρήτρα της ανωτέρας βίας της οποίας κάνουν, την οποία καταχρώνται οι αεροπορικές εταιρείες, ενώ υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός του 2004. Οι επιβάτες είναι θύματα της κατάστασης αυτή τη στιγμή, δεν έχουν καμία εναλλακτική δυνατότητα και επίσης δεν μπορούν ε, να αναλάβουν το οικονομικό κόστος της κατάστασης αυτής. Ε, ε, οι αεροπορικές εταιρείες λένε ότι δεν χρειάζεται να αποζημιώσουν για πτήσεις οι οποίες δεν έγιναν και αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν μάλιστα και ασφάλειες που έχουν οι επιβάτες που τους καλύπτουν σε μερικέ περιπτώσεις ε, όπως για παράδειγμα στην κατάσταση που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες και πιστεύω ότι θα έπρεπε να αποζημιωθούν πλήρως οι επιβάτες για τις ακυρωμένες πτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ. Περίπου 800 εκατομμύρια επιβάτες ε, χρησιμοποιούν ε, εναέριες μεταφορές, 34% ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 40% εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία μας έδειξε ακριβώς πόσο ευάλωτες ε, είναι οι εναέριες μεταφορές στην Ευρώπη. Πάνω από 16.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στην Ευρώπη και ε, πολλοί επιβάτες είναι καθυλωμένοι ε, είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η ασφάλεια των επιβατών και γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα επαναπροώθησης των προώθηση των ε, επιβατών ε, σε άλλες πτήσεις. Αν ένα τέτοιο σύστημα υπήρχε 66% των καθυλωμένων επιβατών ε, εντός ενός κράτους μέλους ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαν φτάσει στον προορισμό τους χρησιμοποιώντας ένα αλλακτικό μέσο μεταφοράς. Και επομένως, πώς μιλούμε για ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και ε, συντονισμένε μεταφορέ εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δεν υπάρχουν κονδύλια για την ανάπτυξη ενό τέτοιου συστήματο, για την εσωτερική ναυσιπλοεία, για παράδειγμα, πρέπει να έχουμε την πολιτική βούληση να συνεχίσει να κινείται η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Γκάλαγκερ. Έχουν γίνει πάρα πολλές δηλώσεις από τον Επίτροπο ε, Κλάους και γίνονται και προσπάθειες από το Συμβούλιο των Υπουργών για να ληφθεί το θέμα. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα μας υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στα χέρια της ε, σύγχρονης τεχνολογίας όσο ε, ποτέ. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα η οποία βρίσκεται σε απόσταση ε, και χωρίζεται από θάλασσα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς νιώσαμε στο πετσί μας τι ακριβώς συμβαίνει. Από χθε το βράδυ θεωρήσαμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλαξε η κατάσταση και ε, ε, οι απαγορεύσεις επεκτάθηκαν για τη μία, μέχρι τη μία σήμερα πάρα πολλοί πεβάτε έχουν ξεμείνει σε διάφορα μέρη όχι μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και η πρώτη μα μέρημνα θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου, να βοηθήσουμε του ανθρώπου οι οποίοι έχουν ε, οικογενειακά προβλήματα, θανάτου στην οικογένεια, οι οποίοι δεν μπορούν να επαναπατριστούν και οι αεροπορικέ εταιρείε δεν θα πρέπει να του αγνοούν και δεν θα πρέπει να του συμπεριφέρονται σαν να είναι ο κάθε ένα ένας τυχαίο επιβάτη. Ε, με χαροποιεί το γεγονός ότι ο Επίτροπος είπε ότι θα υπάρξει μια ομάδα για να αντιμετωπίσει ε, και να συζητήσει το θέμα των επιπτώσεων της κρίσης αυτής. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος της γυροκοντρόλ, όπως προκύπτει και από την κρίση. Διότι ε, η ηφαιστειακή τέφρα, τα ηφαίστεια, δεν ε, σέβονται γεωπολιτικέ και οικονομικές συνέπειε και όρια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια και να ξέρουμε ότι να αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με 27 διαφορετικές λύσεις δεν είναι δυνατόν. Κύριε Γκάλαχερ, πρέπει να σας διακόψω. Τώρα για ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Βίκη Φόρντ. Εκτός μικροφώνου υπόλοιπες δηλώσεις του κυρίου Γκάλαχερ. Κυρία Φρόντ, ευχαριστώ. Η το ηφαιστειακό νέφος ε, δημιούργησε προβλήματα σε χιλιάδες επιβάτες και οικονομικές απώλειες σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοί μας από όλες τις γωνιές της Ευρώπης έχουν εξεμείνει στις χώρες τους αυτή την εβδομάδα και θα πρέπει να πούμε να ευχαριστεί, ένα ευχαριστώ στον Πρόεδρο, ο οποίος συμφώνησε ότι δεν είναι δημοκρατικό να ψηφίσουμε χωρίς αυτούς. Ωστόσο, το ηφαίστειο μας υπενθύμησε ότι εμείς δεν έχουμε τα ενία του πλανήτη και δεν έχουμε και λύσεις για όλα τα προβλήματα είναι σαφές ότι θα πρέπει να κατανοούμε πολύ καλύτερα τι ακριβώς ε, είναι η ηφαιστιακή τέφρα και τι είναι τα ε, ηφαιστειακά αέρια. Επίσης μας υπενθύμησε πόσο εθισμένοι είμαστε στις εναέριες μεταφορές και στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να μειώσουμε αυτή την εξάρτηση. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και να έχουμε προηγουμένα ε, συστήματα για τηλεδιασκέψεις και επίσης συστήματα για βελτίωση των σιδηροδρόμων και επίσης ε, τα περιτά ταξίδια θα πρέπει να μειωθούν. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δώσει το καλά παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Φόρντ. Για δύο λεπτά ο κύριος Μαρινέσκου. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε τα φυσικά φαινόμενα έκτακτου χαρακτήρα, όπως η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία, δυστυχώς δεν μπορούν να προβλεφθούν. Αντίθετα, μπορεί κανεί να πει ότι η αντίδραση όμω σε αυτό το φαινόμενο δεν ήταν επαρκή. Έχουμε την υποχρέωση να αναλύσουμε σε βάθο αυτό που συνέβη και να προετοιμάσουμε αποτελεσματικά μια απάντηση σε περίπτωση επανάληψη αυτού του φαινομένου. Ήταν ανεπαρκή τα όσα έγιναν. Εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεσπάσει το χάο και δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει και ποιοι είναι ακριβώ οι κίνδυνοι. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα κέντρο, ανεξάρτητο κέντρο εποπτεία, άσχετα ποιο θα είναι το κόστο, ώστε οι εμπλεκόμενοι κάνει εταιρείε και επιβάτε να αποκομίσουν τα κέρδη. Βρέθηκαν σε μια κατακαιρματισμένη κατάσταση οι εταιρείε και αυτό δημιουργήσε πολλά προβλήματα για του επιβάτες δεν υπήρξε η δυνατότητα να δοθούν οι σωστοί προσανατολισμοί στους επιβάτες και να δραχθούν τις ευκαιρίες των εναλλακτικών λύσεων. Η μόνη απάντηση είναι η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ε, ουρανού, εναέριου χώρου, ώστε υπό την ευθύνη ενός ενιαίου οργανισμού να μπορέσουμε να δράσουμε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, είχα αναλάβει την εισήγηση για τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εναέριο Χώρο και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν προχωρήσαμε λόγω των αντιδράσεων του Συμβουλίου και αυτό είναι θλιβερό. Επίσης σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφοράς αγαθών τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συναγάγουν τα συμπεράσματα. Η αντίδραση των κρατών μελών δεν ήταν επαρκής και δεν διασφάλισε να υπάρξουν άλλες δυνατότητες μεταφορών. Στην Ευρώπη σήμερα δεν μπορεί να αγοράσει κανείς ένα ε, ε, εισιτήριο σιδηροδρομικής διαδρομής και να μπορέσει να ταξιδέψει με αξιοπρεπή τρόπο. Πρέπει να συντονιστούμε στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό και ο εξυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου είναι μια προτεραιότητα για την οποία γίνεται πολλή λόγο αλλά δεν ακολουθούν πράξει. Ελπίζω ότι θα έχουν μάθει κάτι τα κράτη-μέλη που είναι σημαντικό. Δεν φτάνει να είμαστε προετοιμασμένοι στη χώρα μα, πρέπει όμω να είμαστε προετοιμασμένοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ, κύριε Μαρινέσκου. μισή λεπτό θα είχε ο συνάδελφο Λαμπρινίδη τώρα, παρακαλώ. Πρόεδρε, ο καλό ο καπετάνιο στη φουρτούνα φαίνεται. Στην ηφαιστειακή φουρτούνα που έχει χτυπήσει την Ευρώπη, η Ένωση άργησε να προβλέψει, άργησε να αντιδράσει και άργησε να προλάβει την εξάπλωση των προβλημάτων για του Ευρωπαίου πολίτε όπω αργήσαμε να αντιδράσουμε άλλωστε και στην οικονομική φουρτούνα αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα. δύο είναι οι άξονε τη συζήτησή μα σήμερα. πρώτον όσον αφορά την απαγόρευση πτήσεων και τον συντονισμό προφανώ δεν γίνεται οι εταιρείε να είναι αυτέ οι οποίε σταθμίζουν ρίσκο ζωή και κόστο για αυτέ και αποφασίζουν πότε και πού πετάμε. αυτό είναι θέμα αρμόδιων εθνικών αρχών. το μόνο απόλυτα θετικό επίτευγμα των προηγούμενων ε, ημερών είναι ότι δεν θρυνήσαμε θύματα δεν τα διακινδυνεύσαμε αλλά όμω σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε τα σύνορα τη ευρώπη θα έπρεπε οι εθνικέ αρχέ από την πρώτη στιγμή να συντονιστούν από την πρώτη στιγμή με το eurocontrol με μετεωρολόγου να δουν αν μπορούν να ανοίξουν του διαδρόμου που σήμερα πια λέμε ότι ανοίγουμε και δυστυχώ λέω εγώ μετά από οικονομική πίεση των εταιριών. αυτό με τρομάζει. δεύτερον σε μια τέτοια χαοτική κατάσταση είναι απαράδεκτο ότι αμφισβητήθηκε η εφαρμογή του κανονισμού αποζημίωση των ευρωπαίων επιβατών ο οποίος ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε να ενεργοποιείται αυτόματα. το γνωρίζετε ότι ελάχιστοι εγκλωβισμένοι επιβάτες έχουν διαβεβαίωση σήμερα από τις εταιρείες τους ότι θα πληρωθούν για τις διανυκτερεύσεις; ότι από αυτούς οι περισσότεροι το πέτυχαν επειδή διαπραγματεύτηκαν σκληρά με τις εταιρείες ενώ η πλειοψηφία δεν έχει τίποτα; εδώ το ευρωκοινοβούλιο πιστεύω ότι πρέπει να διερευνήσει τον τρόπο που οι εταιρείε αντέδρασαν σε σχέση με τον κανονισμό και κατά πόσο τα δικαιώματα των επιβατών έγιναν σεβαστά. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. σε ευχαριστούμε κύριε λαμπρινίδη. Δύο λεπτά τώρα ο κύριος Μπέλετ παρακαλώ. Θα eh, eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα προς όλους σας. Είναι μια έκτακτη κατάσταση φυσικά αυτή και σε σχέση με τι εναέριε μεταφορέ, ε, υπέστησαν αυτές ε, πολύ μεγαλύτερο πλήγμα από ότι μετά την 11η ε, Σεπτεμβρίου. Αυτό έδειξε ότι δεν είμαστε εξοπλισμένοι και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση <clears throat> και πάρα πολλοί επιβάτες κατέληξαν σε μια κατάσταση όπου είχαν απομείνει μόνοι και κανένας δεν τους βοήθησε. Κάτι πρέπει λοιπόν να γίνει κύριε Πρόεδρε κύριε Προεδρεύοντα, ένα ευρωπαϊκό έκτακτο πρόγραμμα για έκτακτες ανάγκες και ειδικά τέτοια πρόβλεπτα περιστατικά πρέπει να υπάρχει και να είναι έτοιμο ώστε να δίνονται πληροφορίες και βοήθεια προς τους επιβάτες που έχουν ε, ξεμείνει στα αεροδρόμια και να μπορούν να έχουν τις αναγκαίες φροντίδες για να μπορούν να διανυκτερέσουν. Πρέπει οι ταξιδιώτες αυτές να, να μπορέσουν να βοηθηθούν αυτό πρέπει να δουλέψουμε για να πετύχουμε. Και η Ευρώπη πρέπει πολλά περισσότερα να επενδύσει διασυνοριακά σε δίκτυα ε, τρένων υψηλής ταχύτητας ε, στους σιδηροδρόμους. Είναι αυτό τεράστια σημασία, διότι οι εναέριες μεταφορές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 πρέπει να υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις για το σιδηροδρομικό δίκτυο υπέρ του περιβάλλοντος, υπέρ της απασχόλησης, υπέρ των πολιτών. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Τώρα στη συνέχεια ο κύριος Τζο Λένι παρακαλώ. Ο κύριος Τζο Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και που είναι αρμόδια για τέτοιε φυσικέ καταστροφέ ε, ε, έχει προετοιμάσει μια έκθεση ιδία ε, πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Ο συνάδελφο Ζουάν Φερέρα είναι εισηγητή. Στην επόμενη συνεδρίασή μα θα ψηφίσουμε προς έγκριση αυτή την έκθεση και θα εντάξουμε το σημείο τη έκρηξη του ηφαιστείου με το σύννεφο Στάχτη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να δραστηριοποιηθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Μπορώ να πω συναδέλφους που είπαν ότι είχαμε προετοιμαστεί με αρνητικό τρόπο σε μια τέτοια φυσική καταστροφή. Δόξα τω Θεώ η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πολλές τέτοιες θεομηνίες και καταδείχθηκε παρόλα αυτά ότι υπήρχαν τεράστια ελλείμματα. Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε. Πέντε ημέρες ε, κράτησε μέχρι ότου ένα αεροπλάνο πετάξει για να συλλέξει κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό το νέφος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά η ίδια η πείρα δείχνει ότι δεν τα πήγαμε τόσο καλά, πρέπει να βελτιωθούμε την επόμενη φορά. Αν κάτι κατέδειξε αυτό το σύννεφο στάχτης, είναι η ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη. Ε, οι ε, εθνικές αρχές λέτε επίτροπε ότι έχουν αρμοδιότητες. Αυτό όμως δεν ικανοποιεί τους πολίτες που έχουν υποστεί θυσίε και πλήγματα. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για την προστασία έναντι φυσικών καταστροφών και για φυσικά την ενιαία κοινή πολιτική για τις μεταφορές. Ε, και σε σχέση με αυτές τις δυνατότητες που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας σας ερωτώ πώς δράτεστε τη ευκαιρία για να βελτιωθούν τα πράγματα όσον αφορά τέτοιες καταστάσεις και να είμαστε είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά τώρα παρακαλώ. Εσείς κυρία έχετε τον λόγο. Η κυρία Ντελβό, ευχαριστώ πολύ. Χάος, παραφο... παραλύ... παράλυση, κακοφωνία, αποτυχία. Πάρα πολλέ οι λέξει είναι που μπορούν να περιγράψουν την κατάσταση αυτή και δεν θα επιμείνω σε όλα όσα υπόθηκαν, ε, ειδικότερα όσον αφορά τι οικονομικέ συνέπειε, τι τεράστιε, ε, τι κολοσιαίε, τι άμεσε ή έμεσε για τι αεροπορικέ εταιρείε. Ε, δεν ξέρω μήπω θα έπρεπε να σκεφτούμε την δυνατότητα ενίσχυση των αεροπορικών εταιριών, όμως έχω και κάποιες ανησυχίες για τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής δεδομένου ότι 150.000 άτομα παραμένουν καθυλωμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου, ότι αυξάνεται εκθετικά οι οικονομικές ε, συνέπειες ε, των τη κατάσταση αυτή. Γιατί περιμέναμε πέντε μέρε μέχρι να συνεδριάσουν οι υπουργοί για να αποφασίσουν κάτι και να υπάρχουν διαφορετικέ ζώνε εναέρεια κυκλοφορία. Για ποιο λόγο λοιπόν ε, δεν υπήρξε ε, υπήρξε μεν ε, η τήρηση της πρόληψης, ε, η οποία ήταν η προτεραιότητα, δεδομένου όμως ότι σήμερα εξακολουθεί να είναι ενεργό το ηφαίστειο, ποιες είναι οι επιπλέον εγγυήσεις που λάβαμε για να ανοίξουμε τον εναέριο χώρο που δεν μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Επίσης, ε, ε, υπάρξει ένα, υπάρχει ένα σύστημα ανατροφοδότησης ανά έξι ώρες, αλλά ποιος θα ενημερώνει συνεχώς σε σχέση με την ασφάλεια των ε, διαδρόμων ε, των εναέριων που θα ανοίξουν. Και επίσης, αν αυτό συνεχίσει, αν επιδεινωθεί ή αν ξαναγίνει, που μπορεί και να ξαναγίνει, μήπως χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό των κρατών μελών και συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει πραγματικών δεδομένων, καλύτερο συντονισμός των κρατών μελών σε εξαιρετικέ και έκτακτες περιπτώσεις και επίση συντονισμό για τον επαναπατρισμό όλων αυτών των επιβατών που έχουν ξεμείνει σε διάφορα μέρη και δεν έχουν τρόπο να γυρίσουν. Τώρα οι μεμονωμένες και κρατικές πρωτοβουλίες τι νόημα έχουν. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση μας φέρνει ενώπιον των εθνών μας. Έγιναν συζητήσεις και διακυβερνητικές αποφάσεις οι οποίες δεν επαρκούν και μάλιστα δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στα στατιστικά μοντέλα. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή για να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις και ε, Δεδομένου ότι είχαμε και μια κατάσταση που άφηνε πάρα πολλού χιλιάδε επιβάτε σε κατάσταση ε, απελπισία. Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, να διασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών και αυτού που πετούν και αυτού που βρίσκονται ε, ήδη εν πτήση και όλα αυτά ε, δημιουργήσαν προβλήματα και δημιουργείται και το μεγάλο ερώτημα, αυτό που ρωτάμε πάντα. Τι κάνει η Ευρώπη το, ο Επίτροπος Κάλλας και η Ισπανική Προεδρία προσπάθησαν να εξασφαλίσουν ε, ε, χρόνο ε, και να προσπαθήσουν να έχουν και ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με τον κατάλληλο τρόπο. Δημιουργούνται ερωτήματα φυσικά και θα πρέπει να εφαρμοστούν και τα δικαιώματα των επιωματών. δεν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται διότι δεν ήταν επαρκή τα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν κατεπηγόντω να επαναπατριστούν οι επιβάτε που έχουν ξεμείνει σε διάφορε χώρε τη Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιε κατεπήγοντε καταστάσει. Σε κάποιε περιπτώσει δεν μπορούν τα θεσμικά όργανα να κλείνουν για το Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να δούμε επίση και τι γίνεται με τα τουριστικά θέματα, τα θέματα επιμελητία, τα οποία μόλι προέκυψε η κρίση ε, πλήχθηκαν από όλε τι ε, ε, πλευρέ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή διότι έδρασε και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να ξεφύγουμε από την κρίση. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ε, εναλλακτικό, ένα σύστημα το οποίο θα υποκαθιστά την, ε, τις πτήσεις. Αυτή τη στιγμή ούτε οι σιδηρόδρομοι, ούτε τα οδικά δίκτυα, ούτε οι θαλάσσιες μεταφορές μπόρεσαν να υποστηρίξουν την κατάσταση. Για ένα λεπτό ο κύριος Σαζάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Πράγματι, αντιμετωπίζουμε μια κρίση στις εναέριες μεταφορές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. 80% των αεροδρομίων έχουν κλείσει. Ελπίζω όμως ότι μπορούμε να βγάλουμε κάποια επικοδομητικά συμπεράσματα από την κατάσταση αυτή. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλες τις τις δυνάμεις, ώστε η έκρηξη αυτή του ηφαιστείου να μην οδηγήσει σε πτώχευση αεροπορικών εταιριών. Δεν ξέρω αν αυτό συζητήθηκε στο πλαίσιο της χθεσινής συζήτησης ε, για την ε, κατάσταση, τη νέα αυτή ε, της εναέριας κυκλοφορίας. Και επίσης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που πρέπει βέβαια να εξακολουθούν να ισχύουν. Και επίσης ε, ελπίζουμε ότι τα, οικονομικ... ότι τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν ε, αποτέλεσμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία των ε, επιβατών, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση για τη μεταφορά υγρών στις πτήσεις. Σημαντικό είναι βέβαια να έχουμε προδιαγραφές ασφάλειας, αλλά δεν θα πρέπει να εξαντλούνται όλα εκεί. Πρέπει να σκεφτούμε τους επιβάτες που βρίσκονται σε διάφορα αεροδρόμια καθυλωμένοι. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά διαπιστώνουμε τώρα ότι ο τομέας της αεροπορίας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και ειδικότερα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για όλους όσους δεν μπορούσαν να πάνε στην κηδεία του Πολωνού Προέδρου στην Κρακοβία. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Τελευταίος αγορητής ο κύριος Ένα 1,5 λεπτό θα έχει ο κύριος να παρέμβει παρακαλώ. Ο κύριος Λάιχφελτ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα έλεγα αξιότιμοι συνάδελφοι κύριε Επίτροπε κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο του εφικτού σε αυτή την κρίση και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασαν ικανοποιητικά. Έδρασαν με βάση την αρχή η ασφάλεια πρώτα. Μπορεί κανείς να συζητήσει αν θα έπρεπε να είχαν αναλυθεί κάποια στοιχεία νωρίτερα μπορεί να, ή μπορούσε να είχε γίνει αυτό αλλά καταρχήν αντέδρασαν σωστά οι αρχές αυτό το οποίο όμως πρέπει να συζητήσουμε και πρέπει να προβληματιστούμε επ' αυτού είναι τι θα γίνει με τους πολίτες, με τους επιβάτες που έχουν ξεμείνει, με τους Ευρωπαίους αυτούς. Εχθές μου τηλεφώνησαν τρεις <coughs> μια οικογένεια που βρίσκεται σε ένα αεροδρόμιο και της δόθηκε η πληροφορία ότι στις 29 λέει η επόμενη πτήση. Θα πρέπει δηλαδή να μείνει πάνω από μια εβδομάδα στο αεροδρόμιο. Ή κάποιοι από τη Νέα Υόρκη που είπαν ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο τους ε, επί μία εβδομάδα γιατί οποιαδήποτε στιγμή λέει μπορεί να πάνε να τους πάρουν για να τους πάρουν στο αεροδρόμιο. Ή μια οικογένεια σε ένα ε, νησί που δεν μπορεί να πληρώσει πλέον ε, την παραμονή της ε, εκεί σε αυτό το μέρος και όμως παρόλα αυτά πρέπει να παραμένει εκεί. Είναι πράγματα που πρέπει να μας προβληματίσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σκεφτούμε και να υποβάλουμε λύσεις, προτάσεις για λύσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους πολίτες. Τους Ευρωπαίους μας δεν μπορούμε να τους εγκαταλείψουμε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να μπορέσουν να γυρίσουν σπίτια τους. Ευχαριστώ. Bueno, gracias, Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που είναι οριακή θα έλεγα, γιατί χωρίς αμφιβολία το θέμα το οποίο συζητούμε είναι φυσικά κατεπήγον και πιεστικό για πάρα πολλούς και ιδιαίτερα για τους πολίτες μας και υπάρχει μεγαλύτερο αίτημα να ακολουθήσει η διαδικασία Catch the Eye με την παρέμβαση που θα δίνει τον λόγο πρόεδρος σε όσους τον ζητούν. Έχουμε όμως πάρα πολλούς που ζητούν και έχουμε κάποιους που ζητούν για να παρέμβουν απλά. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 20 που θα παρέμβουν. Όμως παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να παρέμβουν όλοι αν γίνεται αυτό. Και μέχρι να φτάσει κιόλα ο πρόεδρος ο οποίος αποχώρησε και με τοποθέτησε εμένα εδώ να προεδρεύω για να τον αντικαταστήσω. Και έτσι λοιπόν σε σχέση με την διαδικασία αυτή του Catch the Eye δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε μέχρι τελικής πτώσεως. Ο πρώτος ο οποίος θα, θα λάβει τον λόγο είναι ο κύριος Σιλβέστρης ε, από το Λαϊκό Κόμμα, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό θα είναι. Μετά από ένα λεπτό θα κοπεί το μικρόφωνο. Παρακαλώ, ένα λεπτό κύριο Σιλβέστρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τον ε, Υπουργό της Ισπανικής Προεδρίας που έλαβαν το λόγο και συζήτησαν κάποια, είπαν κάποια πράγματα για την κατάσταση η προτεραιότητα φυσικά σε αυτή την κατάσταση ήταν να διασφαλίσουμε ότι ε, υπάρχει ασφάλεια για όλους και αυτό το καταφέραμε. Πρόκειται για ένα φαινόμενο απρόβλεπτο και ε, Χαίρομαι που δεν υπήρχε κανένα αεροπλάνο εν πτήση κατά τη διάρκεια του φαινομένου αυτού. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα της ασφάλειας υπάρχει και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε. Τώρα, το κατά πόσον μπορούσαμε να προλάβουμε τις καταστάσεις, να μπορούσαμε να δράσουμε πιο έγκαιρα και να ανοίξουμε νωρίτερα ε, την περιοχή στην οποία οι πτήσει είναι πιο ασφαλείς λόγω των τεράστιων σημαντικών οικονομικών επιπτάσεων που υπάρχουν για τις εναέριες πτήσεις και τις αεροπορικές εταιρείε, ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή στιγμή. Υπάρχουν χιλιάδε επιβάτε οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μένουν σε ξενοδοχεία. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο, διακόπτει ο πρόεδρο. Έχει το λόγο ο κύριο Ταραμπέλα. Ακούσαμε πάρα πολλούς ειδήμονες του τομέα των μεταφορών και επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στις οικονομικές συνέπειες αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης και της απρόπτης κατάστασης. Υπάρχουν και ανθρώπινες ψυχές βέβαια, τις οποίες ε, επίσης αναφέραμε. Εγώ μιλάω τώρα από πλευράς του καταναλωτή, ε, των επιβατών ε, που έχουν ξεμείνει στα διάφορα αεροδρόμια και δεν μπορούν να γυρίσουν στις χώρες τους. Το ζήτημα είναι ότι έχουν παραμείνει γιατί δεν υπάρχουν και εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε λοιπόν ε, την αναδιατύπωση των οδηγιών που αφορούν ειδικότερα τις εναέριες μεταφορές, ειδικότερα ε, των ε, χαμηλού κόστους πτήσεων, να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου δεν καλύπτονται από τις διάφορες ασφάλειες και από τις αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση ανωτέρας βίας επιβάτες. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Βαλένς σας παρακαλώ έχει τον λόγο. Δεν παρίσταται ο κύριος Βαλένσα. Ο κύριος Μασίπ παρακαλώ. Ναι, εσεί είσαστε εδώ κύριε Βαλένσα. Έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, χωρί να χάσουμε χρόνο να παρέμβετε. Γιατί διαφορετικά θα χάσει ένα συνάδελφο τον χρόνο αυτόν για να παρέμβει ο ίδιο. Ο κύριο Βαλένσα, σα ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή κατάσταση καταδεικνύει απλώς πόσο αδύναμοι είμαστε απέναντι στι δυνάμεις της ε, φύσης. Ακόμα και ως Ευρωπαίοι θα έπρεπε ω Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε καλύτερα διοργανωμένοι και καλύτερα προετοιμασμένοι για μια άμεση απάντηση και αντίδραση σε τέτοιου είδου ε, κατεπήγοντα. Φυσικά είναι δύσκολο να προετοιμαστεί κανεί για κάτι το οποίο ίσω συμβεί ε, με, μετά από ένα διάστημα 150 ετών. Όμω, βλέπουμε ότι για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο είναι ανεπαρκέστατο. Πρέπει να δοθεί απάντηση στο πώ μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα θέματα. Άλλε ερωτήσει που πρέπει να τύχουν απαντήσεων είναι πρώτον, ποιε κρατικέ ενισχύσει θα προβλεφθούν για αυτέ τι εταιρείε ε, που υπέστησαν πλήγματα και κινδυνεύουν τώρα. Φυσικά πολλά μεγάλα κονδύλια θα πρέπει να διατεθούν για να, βελτιωθούν οικονομική, να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Μια άλλη ερώτηση είναι πόσο, πώς θα μπορέσει να προετοιμαστεί μια στρατηγική για να μας προετοιμάσει μακροπρόθεσμα για να αντιδράσουμε σε τέτοια φαινόμενα. Ο επόμενος κύριος Μασίπ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Επίτροπος μίλησε για το παράλογο και το παροχημένο των ε, διαδικασιών. Ας είμαστε λοιπόν συνεπείς. Χάσαμε υπερβολικές ευκαιρίες. Υπερβολικές συνθήκες ε, και ευκαιρίες ε, για να υπάρξει κοινοτική αρμοδιότητα για τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, του τους ευρωπαϊκούς κοινού ουρανούς. Αν δεν, μπορούσαμε, δεν μπορέσαμε να επέμβουμε τουλάχιστον στον ουρανό, τουλάχιστον στην ίδια την γη εδώ σε σχέση με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των επιβατών και ζητώντας ή μεσολαβώντας να υπάρξει χειρία στις ε, συλλογικές συμβάσεις ε, και στις ε, αντιπαραθέσεις όσον αφορά τις μεταφορές. Ελάχιστες, όχι ελάχιστες προϋποθέσεις αλλά μέγιστες δυνατότητες για παροχή υπηρεσιών στις μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σικέρσκι παρακαλώ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στον ευρωπαϊκό τομέα των εναέριων μεταφορών. Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα μετεξελιχθεί σε μια κρίση ευρύτερη του τομέα των ενεργείων μεταφορών. Πρέπει να συναγάγουμε τα συμπεράσματα, τα ορθά σωστά συμπεράσματα από αυτή την κρίση επιτέλους. Και τώρα όσον αφορά την ασφάλεια του τομέα των ε, εναρίων μεταφορών και το θέμα της ε, κινητικότητας. Ε, αυτό είναι η προτεραιότητά μας βέβαια. Επίσης αυτό που χρειαζόμαστε είναι να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφορών θα έχει ένα, μια υφόρα συνιστόσα, μια συνιστόσα υφορίας. Πρέπει οι μεταφορές να μεριμνήσουμε, οι μεταφορές των επιβατών και αγαθών σε σχέση με τις οικονομικές εξελίξεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ε, συγκυρίας οικονομικής κρίσης να μπορέσουν να προαχθούν. Χρειάζεται επίσης η αμοιβαία υποστήριξη ε, εκφράζοντας αλληλεγγύη στις εταιρείες εναέριων μεταφορών. Ο κύριος Μπόρις παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτή η φυσική καταστροφή κατέδειξε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε τις σωστές διαδικασίες και διεργασίες για την αντιμετώπιση έκτακτων τέτοιων περιστατικών όπως αυτή την έκρηξη του ηφαιστείου. Πρώτον θα έπρεπε να συντονίσει τα μέτρα ασφάλειας η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να είναι σε θέση να συντονίσει τις αποφάσεις μεταξύ της όσον αφορά τις εναερίες μεταφορές. Δεν θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Το άλλο θέμα είναι η οικονομική λογοδοσία. Πιστεύω ότι η ασφάλιση έναντι τέτοιων περιπτώσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η επιμελητιακή υποστήριξη για τους επιβάτες εκείνου που έχουν ξεμείνει θα έπρεπε να διασφαλιστεί. Η κινητικότητα όσον αφορά τα τρένα υψηλή ταχύτητας πρέπει να βελτιωθεί επίσης Και τέλος πρέπει να διασφαλίσουμε ότι επιβάτες που έχουν ξεμείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να έχουν τις σωστέ διεργασίες στη διάθεσή του για να βοηθηθούν και να είναι σεβαστά τα δικαιώματά τους. Όλες αυτές οι διεργασίες πρέπει να διασφαλιστούν λοιπόν. Σας ευχαριστώ ο κύριο Αρσένης παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές τις μέρες βιώσαμε μια πρωτόγνωρη αναστάτωση στις ζωέ μας. Το μέσο για το οποίο εξαρτιόμαστε για να μετακινηθούμε από και προς τις περιφέρειές μας, στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο, το αεροπλάνο, δεν ήταν πια διαθέσιμο. Η αναστάτωση ήταν τεράστια χρειάστηκε να πάρουμε τρένα πλοία λεωφορεία να ξοδέψουμε πολύ περισσότερο χρόνο και πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν καν να παρευρεθούν να έρθουν ω εδώ. Όμω αυτό που είδαμε αυτέ τι μέρε είναι ότι δεν εξαρτώμαστε από το αεροπλάνο είδαμε ότι υπάρχουν εναλλακτικά μέσα είδαμε όμω επίσης ότι οι υποδομές για τρένα ε, υπολείπονται αυτή τη στιγμή στην ευρώπη ε, το επίπεδο τη τεχνολογία τη εποχή μα. μπορούμε άραγε να φανταστούμε μια ευρωπαϊκή ένωση με ένα πλήρε δίκτυο γρήγορων τρένων μια ευρώπη όπου όλε οι αποστάσει κάτω των χιλίων χιλιομέτρων θα γίνονται με τρένο και θα χρησιμοποιούμε αεροπλάνο μόνο για τι πιο μακρινέ ε, ε, αποστάσει. οι κλιματικέ επιπτώσει των αεροπορικών πτήσεων στην ευρωπαϊκή ένωση είναι τεράστιε είναι μεγαλύτερε των δηληστηρίων και μεγαλύτερε των εργοστασίων χάλιβα. Ε, αναφορικά με τι μεταφορέ των. 13... σας ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφε. Τώρα θα λάβει τον λόγο η κυρία Άλβαρεθ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η απάντηση που τώρα μπορεί να δοθεί διευκολύνει τη σημερινή κατάσταση αλλά δεν αποφεύγουμε με αυτές τις απαντήσεις ε, κάτι τέτοιο στο μέλλον και θα πρέπει να δραχθούμε της ευκαιρίας ε, αυτή τη στιγμή την εκπόνηση της ε, Λευκής Βίβλου για να συμπεριλάβουμε, να εισαγάγουμε και να θεσπίσουμε τα αναγκαία κοινά μέτρα για να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση που έχουμε αυτή τη στιγμή στις διασυνδέσεις μας σε σχέση με τις εναέριες μεταφορές. Πρέπει να αντισταθμίσουμε αυτές τις διασυνδέσεις με άλλα μέσα, ενισχύοντας τις εναλλακτικέ λύσεις μεταφορών, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο και έχουν τεράστιες ελλείψεις, όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο ή οι ναυτιλιακές μεταφορές. Γι' αυτό και ο κύριος Κάλλας και ο κύριος Γκρό σε σχέση με την εισήγηση αυτής της έκθεσης και σε σχέση με την Επιτροπή ως Επίτροπος, θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την ανάγκη που υπάρχει να ενισχυθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο, το ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπένσεν παρακαλώ θα λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά πράγματα στη σημερινή συζήτηση, αλλά θα πρέπει να δούμε και λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Διότι αυτά τα οποία βιώσαμε θα τα ξαναζήσουμε. Οι ειδικοί στην Ισλανδία λένε ότι δεν είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, θα υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ε, ανοιχτόμυαλοι και να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για μια κατάσταση που θα μπορούσε να προκύψει και στο μέλλον. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και να κάνουμε κάτι προκειμένου η διαλειτουργικότητα να τεθεί σε ε, κίνηση διότι είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ τον κύριο Μπένσεν. Η κυρία Φαζόν έχει το λόγο.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 σε όλους μας σαφές ότι η ασφάλεια των επιβατών πρέπει να βρίσκεται σε ανώτατη προτεραιότητα. Αυτό μας το έδειξε και η ίδια η φύση. Τα αεροπλάνα βρίσκονται καθυλωμένα στο έδαφος, στα αεροδρόμια. Αναμένουν οι επιβάτες στα αεροδρόμια, έχει παραλύσει ο τομέας των μεταφορών, ε, η οικονομία έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα και τεράστιες απώλειες. Φυσικά οι άνθρωποι μπορούν να ε, σκέφτονται, για παράδειγμα όπως οι ότι όταν οι γεωργοί παίρνουν αποζημιώσεις, και εκείνοι, οι επιβάτε δηλαδή, θα πρέπει και εκείνοι να αποζημιωθούν. Κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Αυτό πρέπει να είναι ένα μάθημα για την Ευρώπη. Να υπάρξουν καλύτερε διασυνδέσεις στο δικό δίκτυο, στο σιδηροδρομικό δίκτυο έναντι των ε, εναερίων μεταφορών. Χρειαζόμαστε άλλα μεταφορικά μέσα εναλλακτικών δυνατοτήτων που θα ρηπαίνουν λιγότερο την ατμόσφαιρα και έτσι θα μπορούμε να μετακινούμαστε καλύτερα ως επιβάτε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Τζούντιτ Μέρκε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω ειλικρινή συλληπιτήρια για εκείνους που επλήγησαν από αυτή την κρίση Γίνεται λόγος για κρίση, οικονομική κρίση, ε, κρίση στις μεταφορές, ε, κρίση πιστοτική. Όμως ε, δείχνουν όλα αυτά πόσο ευάλωτη είναι η κοινωνία μας σε σχέση με τα πλήγματα από αυτές τις κρίσεις. Χρειαζόμαστε ένα δίκτυο ασφάλειας. Κάνουμε λόγο για μια, οικογε... για μια κοινωνία που θα είναι δίκαιη και σωστή απέναντι στο περιβάλλον και θα σέβεται το περιβάλλον. Πρέπει να δούμε όμως και άλλες συνιστώσεις. Πολλοί είπαν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν επενδύσεις σε περιβαλλον περιβαλλοντικά φιλικές μεταφορές σε τρένα υψηλή ταχύτητα και δίκτυα υψηλή ταχύτητα, ώστε να μπορούμε να μετακινούμαστε με του σιδηροδρόμου και με τα πλοία. Αυτό είναι καλό για την κοινωνία, καλό για το κλίμα, για το περιβάλλον και για την αηφορία τη κοινωνίας μας. Και αυτό χρειάζεται η κοινωνία μα Πρόεδρο, Σα ευχαριστώ. Κυρία Μέρκε, θα δώσω τον λόγο στην κυρία Μέσνερ και ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη διότι στον κατάλογο που είχα δεν είχα προσέξει ότι η ομάδα στην οποία νίκε ε, έπρεπε να είχε μπορέσει να παρέμει νωρίτερα. Έχετε τον λόγο κυρία Μέσνε, ζητώ συγγνώμη που δεν σας έδωσα τον λόγο προηγούμενο. Αληθεύει ότι ε, οι επιβάτες βρίσκονται σε επίκεντρο σε όλα αυτά. Θέλουμε οι Ευρωπαίοι επιβάτες να μπορούν με ασφάλεια να μεταφέρονται. Ασφάλεια όμως θέλουμε όσον αφορά τον ευρύτερο τομέα των μεταφορών. Χρειαζόμαστε όλο, όλα τα μέσα μεταφορών και τις πτήσεις. Δεν μπορούμε αντικαταστήσουμε τι πτήσει. Έγινε πολλή λόγο για δίκτυα υψηλή ταχύτητα των σιδηροδρόμων. Καλό είναι να έχουμε ε, τέτοιου σιδηροδρόμου υψηλή ε, ταχύτητα. Τι ωφελούν όμω αυτοί οι υψηλή ταχύτητα σιδηρόδρομοι όταν στα σύνορα σταματούν επειδή δεν συνεχίζεται το δίκτυο αυτό σε άλλε χώρε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ένα ευρύτερο πλαίσιο ευρωπαϊκών μεταφορών. Και εδώ το ότι όλα τα κόμματα έχουν εκφραστεί υπέρ του να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλου. Είναι θέμα των κομμάτων στα κράτη-μέλη πολιτικά που τροχοπεδούν πολλά πράγματα. Απευθύνω έκκληση να μεριμνήσετε όλοι ώστε στα κράτη σας, στα κράτη-μέλη μας να υπάρξει πράσινο φω για το άνοιγμα του τομέα των μεταφορών σε όλα τα μέσα μεταφορών στην Ευρώπη. Διότι αν πείσουν τα κόμματά μα γι' αυτό και δώσουν το πράσινο φω, θα έχουμε καλύτερε εξελίξει στο μέλλον. Πρόεδρο σα ευχαριστώ κυρία Μέσνερ. Τώρα η κυρία Κορίνα Κρέτσου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι τελευταίε μέρε μιλάμε πάρα πολύ για τι οικονομικέ απώλειες τι οποίε. Ε, έζησαν ε, τα, οι αεροπορικέ εταιρείες. απόλυε οι οποίε είναι πραγματικότητα, διότι πράγματι πρέπει να συνδράμουμε τι αεροπορικέ εταιρείε, και μάλιστα όσο το δυνατόν περισσότερο ενώπιον αυτή τη κρίση, η οποία προέκυψε από το ηφαίστειο στην Ισλανδία. Κρίση η οποία συνεχίζεται. Το πιο σημαντικό είναι η προστασία των επιβατών, και ε, εδώ υπήρχαν πολλά προβλήματα. Βρίσκονται επιβάτες σε διάφορες χώρες και η αντιμετώπιση δεν είναι κοινή. Εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια ενιαία προσέγγιση, διότι αυτή τη στιγμή οι επιβάτες ε, αντιμετωπίζονται ως πακέτα και τους πάμε από τη μία στην άλλη και περιμένουν να ανοίξουν ένα αέριο χώρο για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η κρίση αυτή που βιώνουμε εδώ και λίγες μέρες δείχνει την αποτυχία της στρατηγικής Λισαβόνας και δεν αφέρθηκε αυτό αρκετά. Ήταν μια στρατηγική που εφαρμόσαμε την τελευταία δεκαετία και μάλιστα η αποτυχία αυτή φάνηκε κατάδυλα με την κρίση αυτή. Φάνηκε πόσο ανίκανη ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονιστεί όταν είδε την κρίση να πλησιάζει και όχι μόνο να προστατεύσει αυτούς που έχουν αποκλειστεί που είναι καθυλωμένοι στα αεροδρόμια αλλά για να μπορέσει να δώσει και μια προοπτική αφήνοντας τις αεροπορικές εταιρείε να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον δοκιμαστικές πτήσεις. Γιατί λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, χρειαζόμαστε περισσότερες κοινοφελείς υπηρεσίες, σε ένα τόσο σημαντικό τομέα όπως είναι οι ενέργειες μεταφορές, γιατί αυτή η απορρίθμιση οδήγησε σε αποτυχία. Ευχαριστώ κύριε Παρνία. Κυρία Φερέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι η κρίση αυτή ήταν απρόσμενη, απροσδόκητη και η αρχή της προφύλαξης έπρεπε να εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα. Αλλά θα πρέπει να αντιλήσουμε και κάποια διδάγματα. Καταρχήν, για πέντε μέρες ε, δεν ακούσαμε ούτε μία στεντόρια και πολιτικά υπεύθυνη φωνή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ακούσαμε αυτή τη φωνή για να προσπίσει τα δικαιώματα των επιβατών, για να διαλευκάνει τα δικαιώματά τους, για να βρει εναλλακτικού τρόπους μεταφοράς και να προβεί σε κάποιο συντονισμό. Το δεύτερο συμπέρασμα που μπορούμε να αντιλήσουμε είναι ότι η διέξοδος ε, από την κρίση δεν θα πρέπει να είναι για τον απλό πολίτη μια διελκυνστίδα μεταξύ συμφερόντων. Θα πρέπει να προσπίσουμε την αρχή της προφύλαξης και τα συμφέροντα των πολιτών. Χρειάζεται να εφαρμόσουμε διαφάνεια και αντικειμενικότητα σε ό,τι αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα εξέλθουμε από αυτή την κρίση στις εναέριες μεταφορές. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό. Διακόπτει ο πρόεδρος την κυρία Φερέιρα. Ο κύριος Γκέρενς είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ο κύριος Γκέμπερ, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, η αρχή της προφύλαξης έχει μετατραπεί σε αρχή ανευθυνότητας, γιατί απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, η αρχή της προφύλαξης ουσιαστικά οδηγεί στην αποποίηση πάσης ευθύνης. Οι θύνοντες δυστυχώ δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους, γιατί είδαμε την πανδημία, τον κίνδυνο για την πανδημία της γρήπης και την έκκληση ε, για μαζικούς εμβολιασμούς πριν καν έχουμε σοβαρή απειλή, πριν καν οποιαδήποτε επιστημονική απόδειξη ότι είναι επικίνδυνη η διέλευση από το σύννεφο της εφεστιακής τάχτης, μας οδήγησε ήδη σε επάυση των αερομεταφορών. Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ αδύναμη και ανίκανη η πολιτική μας και Δυστυχώ φάνηκε η υπερβολική εξάρτησή μα από τι ενέργειε μεταφορέ εξαιτία τη αδυναμία μα να επενδύσουμε στην ανάπτυξη του ε, σιδηροδρομικού δικτύου. Βέβαια, έχουμε τρομερά προβλήματα στι υπεραπόμακρε περιοχέ και ιδιαίτερα στι ενισχυτικέ. Μάλιστα. Τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, Υφυπουργό Λόπε Γκαρίντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. τελικά επιτέχθουν μια συμφωνία στην οποία θα πρέπει να δώσουμε την δέουσα σημασία. Ο βουλευτής Μάικλ Ρεν το ανέφερε σαφέστατα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους μας. Επίσης έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δράση της ενώπιον μιας κρίσης που έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση και έπληξε εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες αλλά και κατοίκους άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έπληξε και την οικονομία, πολλούς σημαντικούς οικονομικούς ε, τομείς. Είδαμε ότι οι αρμόδιοι για το θέμα της, ε, του ανοίγματο των αεροδρομίων ε, συνήλθαν και τελικά οδηγήθηκαν μέσα αυτήν την διάσκεψη, κυρία Σπερώνη, κύριε Φερέιρα, την Παρασκευή μόλις είδαμε ότι υπήρχε μια κατάσταση η οποία ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και παγιωνότανε. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου και με το Eurocontrol εργάστηκαν και την Κυριακή, όπως είπε ο κ. Κάλλας προηγούμενα, υπήρξε ε, παρουσία του κ. Κάλλας της Κομισιόν και εμού προσωπικά δήλωση και τελικά οδηγήθηκαμε στην χθεσινή συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την έκτακτη συνάντηση τη οποία προείδευε ο Υπουργό Ανάπτυξη τη Ισπανία. Ω εκ τούτου λοιπόν ενεργήσαμε. Ενεργήσαμε προκειμένου να καταλήξουμε μια απόφαση σε μια δράση, σε ένα προσανατολισμό και με μια προσέγγιση ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Και σήμερα εφαρμόζονται εφαρμόζεται η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών. Το Ευρωκοντρόλ σήμερα το πρωί από τις 8 έχει προσδιορίσει τέσσερις περιοχές με μια περίμετρο ασφαλείας διευρυμένη όπου δεν θα είναι δυνατόν να γίνονται πτήσεις και υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου θα καταστεί αυτό εφικτό αρκεί να υπάρξει ο παρέτητος συντονισμός ανάμεσα στα κράτη και τις αρχές και θα υπάρξει άνοιγμα των εθέρων και φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί από τις φυσικές και μετρολογικές συνθήκες. Ήδη σήμερα λοιπόν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και αυτό θα συμβεί από εδώ και στο εξή πάντα με την αρχή τη προφύλαξη εγγυόμενη παράλληλα την ασφάλεια. Είδαμε λοιπόν άμεσα ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι αυτή η οποία μας επέτρεψε να λάβουμε μια ισορροπημένη απόφαση. Λάβαμε λοιπόν υπόψη πάρα πολλούς παράγοντες ε, που θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη όταν συμβαίνει κάτι το τόσο έκτακτο όπως αυτό το οποίο ζούμε τις μέρες αυτές. Το μοντέλο αξιολόγησης του κινδύνου είναι πολύ σαφές. Κύριε ε, όταν ε, αναφέρατε αυτό το ζήτημα, θα σα πω ότι το Eurocontrol λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που του παρέχονται από το Λονδίνο. Λαμβάνει υπόψη φυσικά και τις δοκιμαστικέ πτήσει που έγινε. Λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που έρχονται από τους κατασκευαστέ αεροσκαφών. Λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες από την υπηρεσία της κολονίας. Όλα αυτά λοιπόν αξιολογούνται και έτσι είναι ένας πίνακας πολύ σαφής, συγκεκριμένος, όπως αυτό που έχουμε σήμερα απέναντί μας μετά από τις αποφάσεις και τις δηλώσεις των τεχνικών, των επιστημόνων και του Eurocontrol. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη την ασφάλεια που είναι βασικό θεμελιώδες ε, ζήτημα και συμφωνώ με τις παρεμβάσεις που μίλησαν για το ζήτημα αυτό λαμβάνουμε υπόψη τις οικονομικές ε, επιπτώσεις και η Κομισιόν ε, εσύστησε μια ομάδα εργασία ε, προκειμένου την προσεχή εβδομάδα να υποβάλουμε μια έκθεση σχετικά με θέματα που άπτονται τη οικονομία και τι επιρροές αλλά και τα δικαιώματα κυκλοφορίας και κινητικότητας των πολιτών. Ζητώ από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να διευκολύνουν τον επαναπατρισμό των πολιτών και να θέσουν στην υπηρεσία τους όλα τα μέσα επικοινωνίας και μεταφορών έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο στα σπίτια τους να μεταβούν στον προορισμό που επιθυμούν και άρα να εφαρμοστεί η ελεύθερη κυκλοφορία. Για το μέλλον λοιπόν νομίζω ότι με το θέμα αυτό ανοίγει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος ε, όλοι μας μεταξύ αυτών και το Ευρωκοινοβούλιο που αφορούν και το δικαίωμα των ε, επιβατών σε τέτοιες έκτακτες περιστάσεις. Η δημιουργία ενός ε, σχεδίου έκτακτης ανάγκης απαιτεί διαφάνεια όπως είπε η κυρία Βιλμπάου κατά την εφαρμογή και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρξουν διαθροτικές μεταρρυθμίσεις σημαίνει ενίσχυση των μεταφορικών μέσων και δικτύων στην Ευρώπη, ε, ενίσχυση των συνδρομικών μεταφορών. Αυτό είναι στρατηγική σημασία. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διασύνδεση στην Ευρώπη. Δεν δηλαδή, πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη της Ευρώπης οφείλεται στην αύξηση των ε, διασυνδέσεων, των δικτύων, των συνδρομικών δικτύων, των οδικών. Και αυτή η διάρθρωση των δικτύων στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι ότου να υπάρξει μια ολοκλήρωση των υποδομών επικοινωνίας και ιδιαίτερα μέσω των σιδηροδρόμων. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα πολιτικού χαρακτήρα αλλά και συμβολικού συνάμα η βελτίωση λοιπόν αυτών των υποδομών που είναι ένα κεντρικό στόχος για την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Θεωρώ λοιπόν ότι η έκκληση του κ. Ζόβου του για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών από τον κ. Σούλτ, από την κ. Άλβαρη και άλλων νομίζω ότι τίθεται την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χρόνο, διότι αυτή είναι η στιγμή την οποία θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο τη Ισπανικής Προεδρία. Διαδικαστικό. Θα ήθελα να παραταθεί ο χρόνος για τη συζήτηση αυτή, γιατί παρά είναι αυρή αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Γιατί ε, ο κόσμος αντιμετωπίζει για σκουπίδι στις, αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Παρά είμαστε ευγενικοί λοιπόν. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να λάβουν τις πληροφορίες που δικαιούνται. Καταρχήν δεν δίνονται πληροφορίες, ε, μένουν να αβοήθητοι οι επιβάτες ε, εγκαταλειμμένοι στη μοίρα τους και είμαι αγανακτισμένος με την αντίδραση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποτίθεται ότι κόπτονται για τα δικαιώματα των επιβατών τους οποίους αφήνουν να παίρνουν ε, νύχτες ολόκληρες στους σταθμούς και στα αεροδρόμια. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το χρόνο που προβλεπόταν για τη σημερινή συζήτηση και όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων έθιξαν αυτό το ζήτημα δεν έχει μικρόφωνο δυστυχώ, ο Okay. Uh, all this, uh, well, okay. Uh, colleague, sorry, sorry. Uh, all these points were... Όλα αυτά τα θέματα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση στην προηγούμενη συζήτηση, αγαπητέ συνάδελφοι. Λυπούμε, λυπούμε ειλικρινά. Ολοκληρώθηκε ο χρόνο για τη συζήτηση αυτή. Θα ακούσουμε τώρα τον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει μια απάντηση και μετά θα περάσουμε σε ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα. Γιατί περιμένουμε τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μπαρόζο, για τη συζήτηση ενό πολύ βαρισίμαντο θέματο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τι παρατηρήσει σα. Τέσσερι ακόμη παρατηρήσει. Έχω πρώτα απ' όλα βεβαίω το γεγονό αυτό μας κάνει να σκεφτούμε στρατηγικά και οπωσδήποτε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα είναι η διαλειτουργικότητα και η ευελιξία μεταξύ των διαφόρων μορφών μεταφορών και το πώς θα είναι εναλλακτική λύση η σιδηρόδρομη. Και σύντομα θα δούμε την αναδιατύπωση του σιδηροδρομικού πακέτου και τη Λευκή Βίβλο για τις μελλοντικέ μεταφορές. Είναι οπωσδήποτε πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα και χτες το συζητήσαμε και με το Συμβούλιο των Υπουργών. Οπότε είναι σοβαρό αυτό το ζήτημα και βεβαίως το πώς θα περιορίσουμε τις ε, περιτές, ε, την περιττή ανάγκη ταξιδιών. Βεβαίως όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο θα κάνουμε κάποιες προτάσεις με τους συναδέλφους αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γνωρίζετε ότι τα λεφτά δεν έρχονται από το πουθενά και πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σχέση και με τους άλλες επιχειρήσεις. Οπότε πρέπει να, είμαστε, να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση και δεν γίνονται θαύματα τώρα. Για τα δικαιώματα των επιβατών οι κανόνες είναι σαφείς. Με ρωτήσατε ποιοι είναι οι κανόνες και να τους ξαναδούμε. Δεν πρέπει να ξαναδούμε τους κανόνες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγραψε αυτούς τους κανόνες. Είναι πάρα πολύ καλός. Βεβαίω, η εφαρμογή είναι στα χέρια των κρατών μελών και νομίζω πως υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το τι θα κάνουμε για την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Και για το πώς θα επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη, γιατί είναι σαφές το τι πρέπει να γίνει για τις ανησυχίες ε, των επιβατών. Βεβαίως, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που δεν είναι τόσο μεγάλο. Είπαν κάποιοι συνάδελφοι πως ε, έγινε πάρα πολύ αργά, δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Εγώ ήμουν στο Eurocontrol. Ήμουν σε επαφή με τους υπουργούς και εδώ στην αίθουσα έχετε το ίδιο δίλημα που αντιμετώπιζαν και οι ειδικοί και αυτοί που ελάμβαναν τις αποφάσεις. Και αυτό αφορά τους ειδικού και τις αρχές ασφαλείας. Το δίλημα είναι ασφάλεια έναντι ευελιξίας. Είμαστε προετοιμασμένοι για μια έκρηξη ηφαιστείου, αλλά για κάτι το διαφορετικό. Ε, αυτό αναφέρθηκε. Ξέρετε την πτήση της British Airways, ε, της ε, KLM που έπεσε, έπεσε αεροπλάνο της KLM πετώντας κοντά σε ηφαίστειο. Οπότε υπάρχει πραγματικά σοβαρός κίνδυνος και αυτόν έλαβαν υπόψη οι αρχές. Είναι σοβαρός ο κίνδυνος και οι πτήσεις πρέπει να ακυρωθούν. Τώρα έχουμε μία πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση. Την Κυριακή έγιναν οι περισσότερες δοκιμαστικές πτήσεις και είχαμε πληροφορίες στο Eurocontrol όπου συζητήσαμε αυτά τα πράγματα. Οπότε είχαμε δοκιμαστικές πτήσεις. Αλλά τελικά εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη. Έχουμε τον ενιαίο ουρανό, ένα πολλά υποσχόμενο έργο και έχουν συμφωνήσει οι υπουργοί πως είναι σημαντικό για το μέλλον να έχουμε περισσότερο συντονισμό, πως αυτό πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, αυτή, αυτά ήθελα λοιπόν να σας πω. Όσον αφορά την πληροφόρηση, και η Κομισιόν έβγαλε ανακοινώσεις τύπου ήδη από την Πέμπτη. Πέμπτη, πρώτο πράγμα, δικαιώματα επιβατών και ότι θα το δούμε και πολύ σοβαρά. Οπότε πληροφόρηση για τα δικαιώματα επιβατών ήταν άμεση από την Κομισιόν. Και ε, την Κυριακή ξεκίνησε η μεγαλύτερη κάλυψη και χθε βεβαίω ήταν πάρα πολύ μεγάλη όσον αφορά όλα αυτά τα ζητήματα. Οπότε δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση. Έχουμε τρεις-τέσσερις διαφορετικούς ε, τρόπους. Ε, αλλά σας λέω για την οικονομία και τους επιβάτες θα ξαναξεκινήσουν οι πτήσεις ε, και θα φέρουν τους επιβάτες στις χώρες τους ή θα τους πάνε στον προορισμό τους. Οπότε είναι δύσκολη ακόμα η κατάσταση και υπάρχουν συνέπειες που πρέπει να, δούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις ε, παρατηρήσεις σας και οπωσδήποτε θα έχουμε ευκαιρίες να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση που ολοκληρώσαμε για το θέμα αυτό αγαπητοί συνάδελφοι σίγουρα ήταν το πιο σημαντικό θέμα της ολομέλειας αυτής. Και αν μη τι άλλο για αυτή την συζήτηση άξιζε που ήρθαμε στο Στρασβούργο για να ε, το συζητήσουμε, για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Γιατί αυτό περιμένουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτε, να εγγύψουμε στα προβλήματά του. Και αυτό κάναμε σήμερα από το πρωί. Ασχοληθήκαμε με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσω τους 14 ε, επιτρόπους που έλαβαν μέρος στην Ολομέλη αυτή και άκουσαν την πολύ σημαντική αυτή συζήτηση.